Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Θέλω να χαιρετήσω πρώτα απ' όλα τον αντιπρόεδρο Σασολί Βίλαν που ήρθε εδώ σήμερα για να μας μιλήσει για το σχέδιο προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2016. Έχουμε και τον Γενικό Γραμματέα βέβαια μαζί μας. Ήταν ξανά μαζί μας πριν από δύο εβδομάδες για να μας ενημερώσουν για τα πρώτα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον προπολογισμό αυτών του 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόσφατα μάθαμε ότι επεβίωσε ένας ε, συνάδελφός μας, ο κύριος Γιώργος Σταυρακάκης. Ήταν στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και το 2013-2014 ήταν εισηγητής για τον κανονισμό και για το Ταμείο Αλληλεγγύης υπεύθυνο για την συνεργασία με την Επιτροπή Ρέγγι Περιφερειακών Υποθέσεων. Οι εργασίες του αυτές οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές στον κανονισμό. Σκεφτόμαστε λοιπόν τον συνάδελφο αυτό και στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και στους συγγενείς και φίλους του. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε και ένα σεμινάριο προβληματισμού στις 31 Μαρτίου. Πρόκειται για ένα σεμινάριο το οποίο θα αρχίσει νωρίς το πρωί και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική στιγμή αυτό το σεμινάριο στη δράση μας, γιατί θα εξετάσουμε επικριτικά τα όσα τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, θα αναρωτηθούμε για τις επιδόσεις μας. Οι δημόσιες δαπάνες που εμείς εγκρίνουμε είναι μια πραγματική προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη. Και ανταποκρινόμαστε στην πραγματικότητα, στα προβλήματα τα οποία καλούμε θα αναλύσουμε. Μήπως μερικές φορές είμαστε θύματα αδράνειας που μας κάνει να μένουμε πολύ πίσω σε σχέση με τα γεγονότα, με την πραγματικότητα και τις δαπάνες όταν αυτές εκτελούνται. Ιδιαίτερα μάλιστα τώρα που βρισκόμαστε σε παγκοσμιοποίηση. Είμαστε πολύ άριθμοι λοιπόν που θέλουμε να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε αυτά. Σας υπενθυμίζω λοιπόν την ημερομηνία αυτή που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική του σεμιναρίου στις 31 Μαρτίου. Τώρα, έγκριση ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε. Έχουμε επίσης και τα πρακτικά της 26ης Φεβρουαρίου. Τα έχετε. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι από ό,τι βλέπω. Εγκρίνονται συνεπώς. Και έτσι τώρα θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου προπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το οικονομικό έτος 2016. Θα δώσω το λόγο στο Ζεράρ Ντεπρέ, τον εισηγητή μας. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή. Μια που προχωράμε, βέβαια προχωρούν και οι προθεσμίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τους προσανατολισμούς για τον προπολογισμό 2016 πριν από τα τέλη Απριλίου. Περνάει λοιπόν ο καιρός και το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά σφιχτό. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω στους συναδέρφους ότι στην Επιτροπή μας αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καθορίσουμε την θέση μας, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να έχουμε και διαπραγματεύσεις με το Προεδρείο μια από προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2016 θα είναι έτοιμο εφόσον υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στην Επιτροπή Προπολογισμών και το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν λοιπόν θα έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτησή μας εδώ στην Επιτροπή μας, θα έχουμε καταλήξει στις κατευθύνες γραμμές μας, στην τοποθέτησή μας, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την αντιπροσωπεία του Προεδρείου. Το έγγραφο εργασία μου το έχω ήδη παρουσιάσει. Όσοι το διάβασαν λοιπόν δεν θα εκπλαγούν από τις κυρίες κατευθυντήριες γραμμές της έκθεσης αυτής. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μεταξύ των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών που πρέπει να εγκρίνουμε υπάρχει μία που είναι σημαντική και αυτή είναι η προτεραιότητα για τα κονδύλια και για την ενίσχυση του προσωπικού που πρέπει να βασιστεί στην υπευθυνότητα των Ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι συνομοθέτες και που έχουν την ευθύνη ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαχειρίζεται και εκτελεί τα προγράμματα και τα κονδύλια που έχει στη διάθεσή της. Δεύτερον, Στο σημερινό δημοσιονομικό πλαίσιο πολλών χωρών, ξέρετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για να μην αναφερθώ συγκεκριμένα στην πολύ δύσκολη κατάσταση που ζει μια χώρα του νότου της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να έχει μια συμπεριφορά παραδειγματική. Πρέπει δηλαδή να δείξει στο σύνολο της κοινή γνώμης ότι τα κονδύλια τα οποία διαχειρίζεται είναι κονδύλια που είναι αναγκαία και τα οποία δεν έχουν χαρακτήρα οπορτουνιστικό, ούτε πρόκειται για σπατάλες. Έπειτα, για να είναι σαφές για τους συναδέλφους, θέλω να πω επίσης ότι στον προπολογισμό υπάρχουν δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να περιοριστούν. Οι δαπάνε που έχουν να κάνουν με το προσωπικό, για παράδειγμα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί οι δαπάνε αυτέ για το προσωπικό είναι δαπάνες οι οποίες καθορίστηκαν από το ε, καταστατικό που αφορά το προσωπικό. Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με αυτό, αποτελεί όμως μια, ένα σημείο αναφοράς. Έπειτα μην ξεχνάμε ότι κάποιες προσπάθειες που έγιναν να αλλάξουν αυτά καταδικάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μάλιστα με αναδρομικό αποτέλεσμα. Το καταστατικό αυτό λοιπόν προβλέπει κάποιες προσαρμογές περιοδικά για το προσωπικό μας. Αυτό που ονομάζεται upgrading. Όλα αυτά υπάρχουν. Είναι και στο άγγραφο εργασίας μου, αλλά νομίζω ότι η πρότασή μου θα βρει σύμφωνη την Επιτροπή μας και η αύξηση του προβλησμού του Κοινοβουλίου για το 2016 να διατηρηθεί κάτω από το 20% του συνόλου των διοικητικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου λοιπόν του περιθωρίου που είχαμε για τις δημοσιονομικές πρόπτικες, ο στόχος αυτός είναι εφικτός. Θα έλεγα και εύκολα, μάλιστα, με τους στόχους που σας προτείνω. Ο πρώτος λοιπόν να μείνουμε κάτω από το 20% του συνόλου των διοικητικών δαπανών. Δεύτερον, όσον αφορά την αύξηση των δαπανών του προπολογισμού 2016 σε σχέση με το 2015, εδώ έχω μια πρόταση ισορροπημένη πιστεύω. Δηλαδή το ποσοστό αύξησης το 2016 σε σχέση με το 2015 να είναι το αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Πρώτον, εξέλιξη των τρεχουσών δαπανών προσωπικό, συντήρηση, αφαρισμός, αποστολές που έχουμε δεξιά και αριστερά, τρέχουσες δαπάνες λοιπόν. Η αύξηση αυτών των δαπανών το 2016 να διατηρηθεί κάτω από το 2%. Πέρα από το ποσοστό αυτό, προβλέπουμε έκτακτη γρικοδότηση, έκτακτη, για να καλύψουμε τις δαπάνες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Την ασφάλεια των κτηρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή μάλλον δεδομένου ότι αυτές είναι αναγκαίες, έτσι, το ξέρουμε. Υπάρχουν απειλές που υπάρχουν σήμερα και δεν υπήρχαν παλιότερα, οπότε πρέπει να προσαρμοστεί ο εξοπλισμός ε, της ασφαλείας μας, γιατί ο εξοπλισμός που έχουμε τώρα είναι από πριν από 15-20 χρόνια. Συνεπώς, επιγόντως χρειάζεται προσαρμογή και όσον αφορά την κυβέρνηση ασφάλεια. Επίσης, έχω δει διάφορα σημειώματα τα οποία λένε ότι η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχυθούν. Άρα, είπαμε, αύξηση 2016 σε σχέση με το 2015, τρέχουσες δαπάνες κάτω από 2% και έκτακτες δαπάνες για την ασφάλεια. Το Προεδρείο θα ζητήσει, αυτό το συμπέρασμα βγάζω από κάποιες ιδιαίτερες συζητήσεις που είχαμε μέλη του Προεδρείου, θα ζητήσει λοιπόν στις έκτακτες αυτές δαπάνες να προβλέψουμε και την πληρωμή για κάποια κτίρια. Ο Γενικός Γραμματέας φαντάζομαι θα αναφερθεί σε αυτό, δεν θα μιλήσω εγώ περισσότερο γι' αυτό τώρα. Οπότε εγώ δεν μπορώ να κρίνω, η Επιτροπή μας θα αποφασίσει αν θεωρεί ότι είναι δικαιολογημένο το αίτημα αυτό το οποίο θα διατυπωθεί υποθέτω κάποια στιγμή από το Προεδρείο στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που θα έχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Τώρα, Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις προτεραιότητες για το κοινοβουλευτικό έργο. Εδώ προτείνεται να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα της γραμματείας των κοινοβουλευτικών επιτροπών, των ειδικών και ιδιαίτερα στον τομέα του ελέγχου. Ήδη έγινε μεγάλη προσπάθεια τα χρόνια για να βοηθήσουμε τις κοινοβουλευτικές επιτροπές να μπορούν ως συνομοθέτες να δράσουν πιο αποτελεσματικά, ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτικό έλεγχος. Εδώ λοιπόν μένουν διάφορα πράγματα να γίνουν και ο Γενικός Γραμματέας σίγουρα θα προτείνει, θα μας πει τι έχει υπόψη του να προτείνει μάλλον για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Πρόκειται λοιπόν για ενίσχυση της ικανότητας των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ε, είτε με προσωπικό ή μεγαλώνοντάς τες, εν πάση περιπτώσει μάλλον αυτό που χρειάζεται είναι 20 επιπλέον συνεργάτες. Σε σχέση πάντα με την ενίσχυση αυτή του κοινοβουλευτικού έργου, της στήριξης δηλαδή του έργου αυτού, εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε τα πιο δύσκολα ζητήματα προκειμένου να εκπονηθεί ο προπολογισμός 2016. Και αυτό είναι οι αποζημιώσεις γραμματείας οι οποίες δίνονται στους βουλευτές για να πληρώνουν τους διαπιστευμένους τους βοηθούς και άλλους βοηθούς. Ποια είναι τα προβλήματα εδώ. Πρώτον, ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε κάτι που η Επιτροπή μας θα έπρεπε να εγκρίνει. Αντεμνητέντε σεκρεταριά, αποζημίω γραμματεία. Είναι ένα όρο ο οποίο δεν είναι σαφή, γιατί δίνει την εντύπωση ότι παίρνουμε κάποιε αποζημιώσει και εμεί αποφασίζουμε να τι δώσουμε σε ποιον συνεργάτη μα, πώ και τι. Ορισμένοι πιστεύουν ότι επειδή πρόκειται για τέτοια αποζημίωση, αν δεν τη χρησιμοποιήσουμε πλήρω, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και κάπου αλλού. Η ιδέα αυτή, λοιπόν, η ορολογία πιο σωστά που χρησιμοποιούμε δεν είναι κατάλληλη και γι' αυτό θέλω όλοι να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει, ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον άλλο όρο που να είναι πιο ξεκάθαρος και να μην επιτρέπει παρεξηγήσεις και υπονοούμενα. Δεύτερον, δεν επιμένουμε, αλλά κάποιες πολιτικές ομάδες θέλουν αύξηση των δαπανών για το προσωπικό. Άλλες δεν συμφωνούν. Το συνολικό ποσό το, του κονδυλίου για τις δαπάνες του προσωπικού είναι κάτι που δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Τρίτον, πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στους διαπιστευμένους βοηθούς και τους τοπικούς βοηθούς. Δεν θα επανέλθω στα νούμερα, Τα νούμερα όμως μιλάνε από μόνα τους. Η πρότασή μας, συνεπώς, είναι η εξή και θα την βρείτε στο σημείο 14 του σχεδίου με έκθεση. Ζητάμε λοιπόν από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει πρόταση απόφαση στο Προεδρείο, όσο γίνεται πιο γρήγορα, στο Προεδρείο, έτσι, γιατί είναι αρμοδιότητα του Προεδρείου. Και περιμένουμε η τελική αυτή απόφαση να αρχίσει να ισχύει στις αρχές του 2016. Τώρα δεν το λέω σαν απειλή, απλώς υπενθυμίζω ότι η δημοσιονομική διαδικασία μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες κάτω από τις οποίες το Προεδρείο θα αναγκαστεί να τηρήσει τις προθεσμίες που εμείς θέτουμε. Μπορούμε δηλαδή να το κάνουμε αυτό, ώστε οι προθεσμίες που θα θέσουμε να τηρηθούν από το Προεδρείο. Δεύτερο σημείο, σας είπα για την ασφάλεια. Αναφέρθηκα στο Προεδρείο, στο Γενικό Γραμματέα. Μίλησα με τους σκιώδεις εισηγητές τώρα της Επιτροπής μας και ο Γενικός Γραμματέας είναι πολύ σημαντικό που έρχεται να μας παρουσιάσει μια συνολική εκτίμηση, αξιολόγηση των μέτρων που θέλουμε να πάρουμε και για την προστασία των κτηρίων μας, αλλά και για την κυβερνοασφάλεια. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στον προπολογισμό για το 2016. Αν είναι σωστή οι υπολογισμοί μου και για τα δύο αυτά συστήματα ασφάλειας, και για τα κτίρια δηλαδή και για την κυβερνοασφάλεια, μιλάμε για 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Αυτό είναι το ποσό το οποίο θα έπρεπε να προβλεφθεί. Τώρα σε σχέση με αυτά που είπα πριν, για το αίτημα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα υποβάλει το Προεδρείο για προκαταβόλη πρόκειται για το Κόντρα Ντανάουερ του Λουξεμβούργου βασικά, για το κτίριο αυτό. Για το αίτημα λοιπόν αυτό του Προεδρείου η Επιτροπή μας δεν θα μπορέσει να απο... δεν έχει στη διάθεσή της και μια συγκεκριμένη ε, άποψη για την μακροπρόθεσμη στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει το Κοινοβούλιο και δεύτερον για το σύστημα το οικονομικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί όσον αφορά την χρηματοδότηση του κτηρίου αυτού. Και γι' αυτό θα ήθελε ο Γενικός Γραμματέας να μας το εξηγήσει. Τη στρατηγική μεσοπρόθεσμα όσον αφορά τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεύτερον ποιο είναι ο οικονομικό μηχανισμό που σίγουρα, όπως έχω ακούσει τουλάχιστον, είναι ιδιαίτερα περίπλοκος, ποιο είναι αυτό ο μηχανισμό που έχει χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση του κτηρίου ΚΑΤ. Να δούμε μήπως πρέπει να κινητοποιήσουμε και κάποιον άλλο πόρο. Τώρα, όσον αφορά την επικοινωνία, θα ήταν καλό να έχουμε μια εκτίμηση όσον αφορά τα χρήματα που έχει δεσμεύσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τελευταία του προεκλογική εκστρατεία για το κοινό. Δεν λέω πόσο αποτελεσματική ήταν αυτή η εκστρατεία για μας, για το κοινό. Λέω, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Να ξέρω τι αντίκτυπο είχε στην κοινή γνώμη, στον κόσμο. Έπειτα διάφοροι συνάδελφοι μου ζήτησαν και κάτι ακόμα. Διαπιστώθηκε ότι στις Ολομέλειες στο Στρασβούργο πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν να έχουν καλύτερο εξοπλισμό, εικόνα και ήχο για τα κοινωνικά μέσα και άλλα. Φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά ικανοποιητική η κατάσταση, οπότε είναι και αυτό ένα αίτημα που έλαβα εγώ και σας το μεταφέρω. Έρχομαι τώρα στο προσωπικό. Με εξαίρεση τις πολιτικές ομάδες, είπαμε ότι θέλουμε 5% μείωση του προσωπικού. Είναι κάτι που έχει εμφασιστεί στα πλαίσια των ε, δημοσιονομικών προοπτικών. 54 θέσεις λοιπόν θα ελευθερωθούν, είτε με συνταξιδότηση είτε για άλλους λόγους. Σημειώνουμε το αίτημα, χωρίς να μπορούμε να το επικυρώσουμε, γιατί περιμένουμε την ε, έκθεση του Γενικού Γραμματέα όσον αφορά την ασφάλεια, γιατί θέλουμε, είπαμε, παραπάνω προσωπικό για την ασφάλεια. Οπότε, σημειώνουμε την αναγκαιότητα που υπάρχει όσον αφορά την ενίσχυση της γραμματείας των κοινοβουλευτικών επιτροπών. 20 άτομα είπε ο Γενικός Γραμματέας ότι φαίνεται ότι χρειάζονται γι' αυτό. Προηγουμένως θα πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες δυνατότητες μεταφοράς προσωπικού εσωτερικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτοί είναι οι κύριοι προσανατολισμοί, κύριες κατευθυντήρες γραμμές, προς το παρόν τουλάχιστον, που έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου, που έχω την τιμή σήμερα να σας παρουσιάζω. Ευχαριστούμε τον Ζεράρντε Πρέ για την παρουσίασή του, λέει ο Πρόεδρος, όσον αφορά τους προσανατολισμούς του προπολογισμού του Κοινοβουλίου μας. Θα δούμε, σε... μας είπε επίση σε τι πλαίσιο θέλει να γίνει συζήτηση. Υπενθυμίζουμε τις προτεραιότητες. Τώρα, πριν ζητήσω από τους συναδέρφους το λόγο, θα ήθελα να στραφώ προς τον Αντιπρόεδρο Σασόλη να μας πει μήπως θέλει να προσθέσει κάτι. Κύριε Σασόλη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία ανάμεσα στο Προεδρείο, τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον εισηγητή. Βλέπουμε τις βασικές γραμμές του προπολογισμού του 2016 και που είναι δυνατόν να εξοικονομηθούν πόροι και πώς με βέλτιστο τρόπο θα μπορούσε να λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Ζεραρντεπρέ είπε πως για τα ε, τρέχοντα έξοδο θα πρέπει να μην υπερβούμε την αύξηση του 2% και θα υπάρχει μία γραμμή για τα τρέχοντα λειτουργικά αυτά έξοδα και μία ε, ξεχωριστή γραμμή για όλα τα υπόλοιπα και υπάρχουν απρόβλεπτες δαπάνες όπως αυτές που σχετίζονται με την ασφάλεια. Έχουμε 28 διαφορετικά κτίρια που μπορούν να χαρακτηριστούν όλα ως ευπαθή. Για να μην στρατιωτικοποιηθούν όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου θα πρέπει να προβλέψουμε διαθροτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και γι' αυτό χρειάζονται επιπρόσθετοι πόροι. Στα σημεία 16 και 17 ο εισηγητής συνόψισε ε, πάρα πολύ καλά όλες τις νέες προτεραιότητες σε σχέση με την ασφάλεια. Η κυβερνοασφάλεια στο σημείο 18 είναι ένα άλλο ζήτημα όπου διαπιστώνουμε ότι χρειάζονται βασικές παρεμβάσεις και ο εισηγητής εντοπίζει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Η νομοθετική, νομοπαρασκευαστική μηχανή του Κοινοβουλίου θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Παραδείγματο χάρη γραμματιακή υποστήριξη για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση. Η πράξη κατεξουσιοδότηση είναι ε, το νομοθετικό μας έργο. Είναι καθήκον μας. Εάν δεν θέλουμε να παρατηθούμε αυτό το ρόλο, το βασικό ρόλο του συνομοθέτη, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε το ρόλο μας. υπάρχουν περίπου 400 ε, πράξεις ε, κατεξουσιοδότηση που ε, εκδίδονται ετησίως. Πρόκειται για, ξαναλέω, για νόμο παρασκευαστικό έργο. Συμφωνούμε απολύτως με τα σημεία 26 και 27 ε, περί αυτών των αυξήσεων. Τώρα, Ας περάσουμε στα ευαίσθητα, πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα για την εξοικονόμηση των πόρων. Έχουν συμφωνηθεί ε, ήδη κάποια πράγματα το 2015 και οφείλουμε να θέσουμε εφικτούς στόχους όπως ε, και πάλι σωστά μας είπε ο εισηγητής το περιθώριο 0,5% που έχουμε ανάμεσα στην ε, στον προϋπολογισμό και στην εκτέλεσή του 14,4 εκατομμύρια ε, τόκων ε, που μας επιτρέπουν να κάνουμε μια σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε λοιπόν το 0,5% το περιθώριο που έχουμε. Όπως είπε ο κύριος Ντεπρέ, θα πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρήσουμε την μείωση των εξόδων προσωπικού ε, κατά 5% που προβλέπεται μέχρι το 2020 προβλέπεται ε, εξοικονόμηση 1.800.000 ευρώ με την ε, μείωση κατά 57 των διαθέσιμων θέσεων, οργανικών θέσεων. Ε, σε σχέση με την αποζημίωση για τη γραμματιακή δουλειά έχουμε τοποθετηθεί Νομίζω ότι είναι αμφίσιμος όρος και δημιουργεί παρανοήσεις. Πρόκειται για χρήματα που διοχετεύονται ουσιαστικά στην κοινοβουλευτική εργασία. Ας προσδιορίσουμε επακριβέστερα περί τίνος πρόκειται. Δεν πρόκειται για αποζημιώσεις, πρόκειται για ένα ταμείο από το οποίο αντλούνται κονδύλια για την κοινοβουλευτική εργασία. Και ξέρετε πως σε όλες τις πολιτικές ομάδες έχει ξεκινήσει μια σχετική συζήτηση και θα συνεχιστεί δεδομένου και του πολιτικού αντικτύπου που μπορεί να υπάρξει στην κοινή γνώμη. Έχει αρχίσει λοιπόν η συζήτηση, συνεχίζεται σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Είναι μάλλον αποκλίνουσες οι απόψεις προς το παρόν. Ε, νομίζω ότι εξυπηρετούμε τους ίδιους οικονομικούς ε, στόχους, θα πρέπει να συμφωνήσουμε και σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν βουλευτές ε, που έχουν δεκάδες ε, ντόπιου βοηθούς όπως ονομάζονται ε, και άλλοι που δεν έχουν βοηθούς ούτε στο Στρασβούργο ούτε στις Βρυξέλλες. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, θα πρέπει να προβούμε στις απαιτούμες μεταρρυθμίσεις για το κεφάλαιο ε, των διατάξεων που διέπουν τη δουλειά των βοηθών, εξασφαλίζοντας την αξιοπρεπία στην εργασία, αλλά μη δημιουργώντας ταυτόχρονα και την πλημελή εντύπωση πως ε, αυτή οι βοηθοί δεν ε, επιδίδονται σε κοινοβουλευτικό έργο. Χρειάζεται λοιπόν μία ισορροπία ανάμεσα στους διαπιστευμένους και τους ντόπιου βοηθούς. Ε, στο σημείο 14 ο κύριος Ντεπρέ ε, πραγματεύεται αυτό το ζήτημα και είμαι σίγουρος ότι το Προεδρείο θα υποστηρίξει και θα προωθήσει τη διατύπωση που έχει επιλέξει ο κύριος Ντεπρέ στο σημείο 14. Δεδομένου του ότι θα καταθέσουμε μια πρόταση που φυσικά σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία όμως θα δημοσιευτεί, θα εξεταστεί από τους πολίτες, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο ώστε να δείξουμε ότι θα προβούμε σε εξοικονόμηση πόρων. Ευχαριστούμε κύριε Σασόλη, κύριος Βίλαντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. συμφωνώ πρώτα με τις ευχαριστίες του κύριου Σασόλη προς τον εισηγητή. Στην παράγραφο του 10 χωρίζει δύο πράγματα ο εισηγητής. Αφενός τα τρέχοντα και αφετέρου τις έξτρα δαπάνες που θα πληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει τα project των παρελθόντων ετών. Έχουμε πάλι πρόσθετες επιβαρύνσεις να αντιμετωπίσουμε και είναι αδιαμφισβήτητο και στο Προεδρείο ότι το θέμα της ασφάλειας και για να το πω με τους δύσκολο να μεταφραστούν στα ελληνικά όρους safety και security, δηλαδή είναι και τα δύο που είναι σημαντικά. Θα ήθελα λοιπόν και μέσα στη γερμανική μετάφραση όπου υπάρχει το ίδιο πρόβλημα μετάφρασης να γίνει διάκριση ανάμεσα σε safety και security. Το ίδιο για την cyber security. Για τη cyber security πιστεύω ότι η συνολική προσέγγιση στην ασφάλεια ασφαλώς αναφέρεται στα, στα κτίρια και χρειαζόμαστε να δούμε και πού προσεγγίζει και πού τέμνει η κυβερνητική ασφάλεια την φυσική ασφάλεια κτηρίων και προσώπων. Βεβαίω αυτά συνεπάγονται κόστος. Ήμουν και αρμόδιος για τον τομέα high-tech τα τελευταία πέντε χρόνια, επομένω γνωρίζω για ποιο πράγμα μιλώ. Έχουμε βέβαια την εσωτερικοποίηση της ασφάλειας ήδη πίσω μας, την έχουμε κάνει ήδη. Έχουμε όμως ακόμη Βρισκόμαστε μάλλον σε επίπεδο κίτρινο των επιπέδων ασφάλειας. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε, αν θα χρειαστεί να έχουμε αστυνομικές δυνάμεις μπροστά από το κτίριο ή και μέσα, με στολή ή με πολιτικά, οπλισμένους ή όχι. Αυτά θα έχουν βεβαίως ξεκάθαρες επιπτώσεις και στο κόστος του προσωπικού. Αν κάνω τη σύγκριση με τη γερμανική Bundestag, όπου είναι βεβαίω πολύ διαφορετικές οι κατηγορίες εκεί και οι δομέ, είμαι πεισμένο ωστόσο ότι για κάποιο διάστημα, τουλάχιστον 6 μήνες ή έω 9 μήνες, θα χρειαστούμε και απ' έξω παροχή συμβουλών. Δεν έχουμε όλη την τεχνογνωσία που μας είναι αναγκαία. Θα χρειαστούμε λοιπόν και λύσεις που να έρθουν απ' έξω, που να προσαρμόζοντας τόσο στην πραγματικότητα. Έχουμε και κάτι το οποίο θα ξεπεράσει και το 2016, άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και μεσοπρόθεσμα, να τα προβλέψουμε δηλαδή και να λάβουμε τις σχετικές δημοσιονομικές αποφάσεις και για τα έτη 16 και 17. Έρχομαι τώρα ε, λίγο στο πρώτο μέρος της παραγράφου 10 για την αντιμετώπιση του κόστους των υποχρώσεων. Όπως είπε και ο κύριος Ντεπρέ, μένει το θέμα της στήριξης του έργου των βουλευτών με επαρκές προσωπικό. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην Ευρώπη της Λισαβόνας, που σημαίνει πολλή δουλειά από πλευράς κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Και το ερώτημα δεν είναι εδώ ποιοι δουλεύουν και ποιοι δουλεύουν, αλλά ποιοι δουλεύουν καλά και αν δουλεύουν όλοι καλά. Ο Χρυσοθύρας καταφέρνει και βρίσκει τους, τα ψήγματα χρυσού μέσα στην άμμο λόγω του διαφορετικού βάρους που έχουν τα ψήγματα του χρυσού. Εμείς κάνοντας τη μεταφορά στο έργο του βουλευτού πώς θα το κάνουμε. Εμείς δεν θέλουμε ως ευρωβουλευτές μοναχά να επιφορτήσουμε τις κοινοβουλευτικές επιτροπές με την ανάγνωση των κειμένων. Αν δεν θέλουμε μόνο οι πολιτικές ομάδες και βέβαια και οι σύμβουλοι να φορτωθούν περισσότερη δουλειά, να ασχοληθούν δηλαδή με τα πράγματα αυτά και να μας τα ετοιμάζουν, μασημένα δηλαδή να μας τα δίνουν, θα πρέπει και οι βουλευτές να μπορούν να παρακολουθούν τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και να μπορούν να κάνουν και την επεξεργασία των κειμένων που περιέχουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Αυτό έχει κάποιες συγκεκριμένε επιπτώσεις. Και για τις γραμματείες τώρα έχω και κάποιες αμφιβολίες εάν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες με τη μαγική λέξη redeployment Βεβαίω έχει αφήσει αρκετά αόριστες διατυπώσεις του ο εισηγητής έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να ε, προσθέσουμε και άλλα πράγματα. Τώρα, θα κλείσουμε τα κενά σιγά σιγά. Καθένας ευρωβουλευτής λοιπόν να μπορεί να έχει και ένα τρίτο χώρο γραφείου ώστε το ερώτημα αν θα χωράνε επιτέλους οι συνεργάτες του ή όχι να λυθεί. Θα εξετάσουμε και από την άποψη του προγραμματισμού των εργασιών του Ευρωκοινοβουλίου έτσι ώστε η δουλειά των βουλευτών να, γίνει και αυτή πιο ευέλικτη και με τον τρόπο αυτό και προς τα έξω δηλαδή αλλά και προς το εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Ορισμένα πράγματα πεντάσσονται ακόμη στο πακέτο, τα είπε ο κύριος Ντεπρέ με τους τοπικούς και διαπιστευμένους συνεργάτες των βουλευτών. Το Κοινοβούλιο εντάσσεται στο πακέτο αυτό με όλες τις υπηρεσίες του, οι πολιτικές ομάδες επίσης και τι γίνεται με τους ευρωβουλευτές τελικά και σε ποιο βαθμό θα βελτιωθεί η θέση των ευρωβουλευτών μέσω της στήριξης των γραμματιών τους. Δεν παραμένουμε μόνο στη λέξη επίδομα, πρέπει να δούμε ορισμένε ομάδες έχουν πει ποιες είναι οι θέσεις τους. Από ορισμένες άλλες πολιτικές ομάδες ακόμα δεν έχουμε τελική θέση. Οφείλω να πω ότι για μια τετραετία έχουμε το επίδομα γραμματείας παγωμένο. Υπήρχε και ένα τεχνικό αποτέλεσμα μιας δικαστικής αποφάσεως. Εάν είχε γίνει μόνο η αύξηση με το ποσοστό με το οποίο αναπτύσσεται ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν είχαμε χρησιμοποιήσει αυτό το ποσοστό δηλαδή, θα, ήταν, θα είχε επιτευχθεί τώρα βελτίωση και του αριθμού των συνεργατών μας και της αμοιβή τους που είναι γύρω στα 1000 ευρώ. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι θεραπεία περιπτώσεων που κατά τη γνώμη μου έχουν γίνει, όπου κατά τη γνώμη μου μάλλον έχουν γίνει σφάλματα στο παρελθόν. Αυτό που θα έρθει τώρα και θα πει εγώ είμαι το φως, εγώ θα τα κάνω όλα μόνος μου, κανένας δεν εμποδίζεται να προσφύγει στο επίδομα γραμματείας. Εάν δεν το χρησιμοποιήσει επανέρχεται στο Ταμείο του Κοινοβουλίου στο τέλος του έτους. Τώρα κάνουμε εξοικονομήσεις και στο χαρτί και στους διερμηνείς. Αυτά όλα αρκούν ώστε τα μερίσματα που θα επιτύχουμε να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αλλού. αλλά νομίζω ότι ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα. Όταν μιλούμε για αποτελεσματικότητα της εργασίας ορισμένες παραγράφους του κειμένου όπως, 15, όπως 5, 16 και 17, αυτά μου θυμίζουν λίγο κάτι αυτή την ε, κότα που κάνει τα χρυσά αυγά. Πώς να το πω. Νομίζω δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ωραιότατες μεταφορές που κάνετε, Πρόεδρε. Πριν από δύο εβδομάδες σας είχαμε μαζί μας, κύριε Γενική Γραμματέα. Έχετε επιπλέον σχόλια πριν δώσω το λόγο στους συναδέρφους δηλαδή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Κύριε Πρόεδρε. Είχα την ευκαιρία προεβδομάδων να σας αναπτύξω τις guidelines, δηλαδή τη γενική κατεύθυνση. Αυτό βέβαια πριν να έχουμε συγκεκριμένα νούμερα. Τώρα το Προεδρείο έχει συζητήσει τα προκαταρκτικά σχέδια των εκτιμήσεων Επομένως μπορούμε να επανέλθουμε τώρα και να σας υποβάλουμε συγκεκριμένα νούμερα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ορισμένα από τα βασικότερα στοιχεία που είναι σημαντικά για τη συζήτησή μας. Πρώτα για τον ρυθμό αύξησης. Όλοι γνωρίζετε ότι παραδοσιακά το Κοινοβούλιο ζητεί 20% του τίτλου 5 των διοικητικών δαπανών του προϋπολογισμού για λογαριασμό του. Αν το πράξουμε αυτό και φέτος, θα δικαιολογήσουμε αύξηση του προϋπολογισμού μας κατά 5,6%. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο δικό τους πολιετή σχεδιασμό έχουν προβλέψει ρυθμό αύξησης των διοικητικών δαπανών. Αν ακολουθήσουμε τη δική τους γραμμή μπορούμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό κατά 4,5%. Αυτό που σας προτείνουμε δεν είναι ούτε το 5,6 ούτε το 4,5%. Προτείνουμε 3,09. Άρα ήδη το Προεδρείο παραμένει σαφώς κάτω από αυτό που θα ήταν δυνατό υπό τον τίτλο 5, αλλά και κάτω από το επίπεδο που προβλέπουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων με την απόφασή τους για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο διεξαγάγαμε ήδη τη συζήτηση με τον εισηγητή. Ο εισηγητής θεωρεί ότι το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι γύρω στα 2%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά γύρω στο 2%. Μας επιφόρτησε ο πρόεδρός μας λοιπόν να ψάξουμε να βρούμε μια λύση που θα κείται γύρω, μάλλον ανάμεσα στο 2 με 3%. Εάν το πράξουμε αυτό θα χρειαστεί να εντοπίσουμε το μίσο που μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις. Μου έχει δώσει την εντολή ο Πρόεδρος αυτό να πράξω, να ψάξω να βρω έξτρα σημεία εξοικονόμησης και η συζήτηση που θα γίνει θα είναι αυτή, δηλαδή τι είδους εξοικονομήσεις μπορούμε ακόμα να εντοπίσουμε στον προϋπολογισμό ώστε να καταλήξουμε σε ένα ρυθμό αύξησης που να μπορεί να γίνει αποδεκτός και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και από το Προεδρείο. Το οποίο Προεδρείο έχει επισημάνει το γεγονός ότι για το 2016 οι δαπάνες θα είναι μεγαλύτερες για την κατασκευή του κτηρίου Conrad Adenauer στο Λουξεμβούργο. Η δαπάνη που θα πρέπει να αναμένουμε είναι της τάξης των 117 εκατομμυρίων ευρώ. Για την ώρα δεν προβλέπεται στο προϋπολογισμό συμβολή στην δαπάνη αυτή. Άρα το ποσό θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με, με λήψη πίστοσης, με δάνειο δηλαδή. Από την άλλη μεριά, αν χρησιμοποιήσουμε όλο το χώρο που δίνει ο τίτλος 5 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 46 εκατομμύρια για να χρηματοδοτήσουμε την κατασκευή του κτίριου Conrad Adenauer, το οποίο για τα επόμενα 15 χρόνια θα εξοικονομήσει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ υπέρ του Κοινοβουλίου και άλλα του φορολογουμένου. Δεν προτείνει αυτή τη στιγμή το Προεδρείο κάτι τέτοιο. Το Προεδρείο προτείνει να διεξαχθεί διάλογος μεταξύ Προεδρείου και Επιτροπής Προϋπολογισμών να δούμε αν μπορούμε να μειώσουμε την επιβάρυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επομένως και των φορολογουμένων με το ε, ποσό αυτό των 15 εκατομμυρίων. Τρίτο, η συζήτηση για τους ε, συνεργάτες των βουλευτών. Αυτή η συζήτηση εξελίσσεται προς την κατεύθυνση που λέει ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μοναχά ένα θέμα, δηλαδή ποιο είναι το ορθό ποσόν και ποια αύξηση θα πρέπει να προβλεφθεί, αλλά να προβλέψουμε και έναν αριθμό μέτρων που σιγά σιγά θα συνδυαστούν και θα οδηγήσουν σε μια μεταρρύθμιση του συστήματος. Μπορώ νομίζω να πω ότι η πλειοψηφία των μελών του Προεδρείου θεωρεί ότι το ποσό θα πρέπει να αυξηθεί και ότι αυτό θα πρέπει να γίνει το 2016. Σωστό είναι επίσης να πω επίσης ότι δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα για το ακριβές ποσό. Υπάρχει συμφωνία ωστόσο ότι ό,τι αποφασίσουμε εδώ θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα. Συχνά διαβάζουμε στον τύπο ότι πρόκειται για έξτρα ποσόν που τίθεται στη διάθεση των μελών, των βουλευτών δηλαδή, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό προορίζεται για την κάλυψη δαπανών, ιδίω βεβαίω ε, συνεργατών, βοηθών, αλλά ιδίω και για την αγορά τεχνογνωσία. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί μέσα στη διαδικασία του προϋπολογισμού ποιο είναι ο σκοπός της δαπάνη. Δεν είναι δηλαδή ένα ακόμη ποσό το οποίο καταλήγει στου βουλευτέ, αλλά είναι δαπάνη προσωπικού. Τρίτο θέμα που πρέπει να συζητηθεί και μου φάνηκε ότι τη Δευτέρα διαμορφωνόταν συνένεση στο Προεδρείο αλλά και συμφωνία με τον εισηγητή είναι ότι εν μέρη βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου σημειώνεται μια μεγάλη έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα σε πρόσωπα που προσλαμβάνονται ως τοπικοί συνεργάτες και στην υποστήριξη που έχουν για το βασικό νομοθετικό του έργο στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο οι Ευρωβουλευτές. Στην διαδικασία χορήγησης απαλλαγής για το 2013 χρειάστηκε να αναφέρω ότι σε ορισμένες χώρες μέλη έχουν φτάσει σε υψηλούς διψήφιους αριθμούς οι συνεργάτες, ενώ στις Βρυξέλλες ισχύει μονάχα το όριο των τριών και μόνο με έξτρα άδεια μπορούν να φτάσουν στους τέσσερις. Αυτή η ισορροπία βεβαίως είναι στρεβλή. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη των Ευρωβουλευτών για το νομοθετικό του έργο και από την άλλη μεριά χρειάζονται βέβαια και κάποιοι περιορισμοί όπου τα πράγματα έχουν παραγίνει όσον αφορά τον αριθμό των τοπικών, των εθνικών συνεργατών δηλαδή. Χρειάζεται κάποια ισορροπία λοιπόν στη στήριξη του έργου στις χώρες και στις Βρυξέλλες. Ένα τέταρτο θέμα που αναφάνηκε στις συζητήσεις του Προεδρείου είναι ότι η σύσταση που έγινε από την ομάδα Ροτ Μπέρεντ για τα επίπεδα αμοιβών των συνεργατών στις χώρες μέλη επιτρέπουν σε κάποιες χώρες μέλη όπως βεβαίω στη Ρουμανία αλλά εν μέρει και στην Πολωνία όπου η μισθή είναι πολύ χαμηλή οδηγούνται εκεί σε καταστάσεις που είναι υπερβολικά περιοριστικές για τις επιλογές των βουλευτών και οδηγούνται και σε άδικες προσεγγίσεις. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναδούμε τους κανόνες αυτούς έτσι ώστε να υπάρχει επαρκή στήριξη στις χώρες μέλη εκείνες όπου είναι πολύ χαμηλές οι αμοιβέ, γιατί και αυτοί οι συνεργάτες αναμένεται από τους εργοδότες τους να γνωρίζουν πολλές γλώσσες, να έχουν καλή ε, ε, μόρφωση, παιδεία και βεβαίως να μπορούν οι βουλευτές να πληρώνουν ένα αξιοπρεπή μισθό. Αυτό λοιπόν που εξετάζει σήμερα το Προεδρείο δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο για μια ενδεχόμενη αύξηση των ποσών που θα είναι διαθέσιμα για την πρόσληψη συνεργατών, εξετάζει ένα συνολικό πακέτο για την αντιμετώπιση του θέματος και για την αντιμετώπιση ορισμένων ε, πραγμάτων που έχουν πάρει μια λάθος πορεία. Τώρα, για την ασφάλεια. Το Προεδρείο έχει λάβει επιπροσθέτως ορισμένες αποφάσεις την περασμένη Δευτέρα, αλλά μπορούμε τώρα να περιγράψουμε με καλύτερο τρόπο ποια μέτρα προβλέπονται πρώτα και αμέσως, δηλαδή το 2015 θα αλλάξουμε την διαμόρφωση των εισόδων των κτίριων εδώ στις Βρυξέλλες, ιδίω της οδού Βίρτς, αλλά και της οδού Λουξεμβούργου, της πλατείας Λουξεμβούργου, με δύο σκοπούς ιδίως. Πρώτα, εάν υπάρξει απόπειρα εισόδου στα κτίρια μας με, από πρόσωπα τα οποία δεν επιτρέπεται να εισέλθουν. Θα πρέπει τεχνικά να έχουμε τη δυνατότητα να τους αποκρούσουμε. Δεν θα είναι δυνατόν δηλαδή απλά να περάσουν. Άρα πρέπει να φτιάξουμε μια ζώνη προστασίας όπου μπορούν τα πρόσωπα αυτά να αναχαιτιστούν. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι γυάλινες αυτές πόρτες δεν θα, είναι, δεν πρέπει να, είναι, να φτάνουν μόνο με στο μισό ύψος του ανθρώπου, αλλά να είναι αρκετό ύψος ώστε να μην μπορεί κάποιος να μπει παρά την αντίσταση των φρουρών μας. Αυτό θα πρέπει να γίνει με απόλυτα σύγχρονα μέσα και γι' αυτό θα θέλουμε να ακολουθήσουμε το πρότυπο της ε, υπηρεσία εξωτερική δράση που είναι η τελευταία που έχει οθετήσει τα μέτρα αυτά ασφάλεια, ε, τα πιο σύγχρονα δηλαδή. Επίση, σε ορισμένου ευαίσθητου τομεί θα πρέπει η προστατευσιμότητα μέσω γυαλιού θα πρέπει να ενισχυθεί. Δηλαδή το γυαλί αυτό θα πρέπει να είναι αλεξίσφαιρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν τα τζάμια αυτά. Ίσως αρκεί να προσθεθεί ένα έξτρα επίπεδο. Άρα πάντως τα τζάμια σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και σε ευαίσθητα σημεία θα πρέπει να είναι αλεξίσφαιρα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σχετικά σύντομα και μέσα στο 2015. Αυτό ενδέχεται να χρειαστεί προκαταβολική δέσμευση και έγκριση κάποιων δαπανών, front loading δηλαδή, γιατί εκεί χρειάζεται να φροντίσουμε για την επαρκή προστασία μας σύντομα και να μην περιμένουμε να περάσει ο χρόνος. Είναι σημαντικό επίσης όλα τα προγράμματα ε, τεχνολογίας της πληροφορικής να μπορούν να διαλέγονται συνεχώς. Αν βρεθείτε σε κρίση δεν θέλετε να έχετε διαφορετικά συστήματα τα οποία να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνδιαλέγονται ταχύτατα. Κάτι λοιπόν το οποίο επίσης πρέπει να επιτύχουμε σχετικά σύντομα. Το Προεδρείο αποφάσισε επίσης την προηγουμένη Δευτέρα ότι θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τα badge, δηλαδή τις άδειες εισόδου. Έχουν αρχίσει τώρα να είναι απειρχαιωμένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει αλλάξει τις δικές της ταυτότητες. Θα ακολουθήσουμε το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν, της Κομισιόν, που σημαίνει ότι θα πρέπει να διαθέτουμε περισσότερες πληροφορίες, γιατί οι ταυτότητες, οι, οι άδειες εισόδου που έχουμε τώρα εύκολα μπορούν να παραχαραχθούν. Ο πέμπτος τομέας είναι cyber security. Δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες αποφάσεις εδώ. Θα χρειαστεί το Προεδρείο να εγγύψει σε θέματα όπως κρυπτογράφηση ηλεκτρονικών ταχυδρομείων και άλλα σχετικά. Έρχομαι τώρα στο πέμπτο σχόλιο μάλλον και αυτό αναφέρεται σε πράξεις κατεξουσιοδότηση ή εκτελεστικές. Αναμένουμε όγκους τέτοιων πράξεων. Ο νέος τομέας θα είναι κυρίως στην Οικονομική Επιτροπή χρηματοδοτικοί κανονισμοί. Ούτως ή άλλως είχε υπάρξει μέγα όγκος εργασίας και στην προηγούμενη θητεία. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι σχετικές επιπτώσεις θα φτάσουν στο Κοινοβούλιο υπό την μορφή σχεδίων εκτελεστικών και κατεξουσιοδότηση πράξεων. Έχει κρίσιμη σημασία να μπορούμε και να τις ελέγξουμε και να επιτρέψουμε στους βουλευτές να στοχεύσουν στα πιο σημαντικά και ευαίσθητα θέματα. Διότι αυτές η πράξη κατά εξουσιοδότηση είναι νομοθετικές πράξεις και το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να πει όχι. Δεν μπορεί να έρθει μετά το Κοινοβούλιο και να πει «Α, δεν πρόλαβα, δεν ήξερα, δεν είδα». Όταν οι πολίτες διαμαρτύρονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ δεν θυμούμαι να διαμαρτύρονται για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Συνήθως διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις νομοθετικών πράξεων εκτελεστικών ή κατεξουσιοδότησης. Δηλαδή πολύ λεπτομερή θέματα. Και το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις πράξεις αυτές. Και γι' αυτό πρότεινα στο Προεδρείο και το στήριξε αυτό το Προεδρείο, καθώς επίσης και ο εισηγητής, στην πλέον θυγόμενη επιτροπή, είμαστε στις πλέον θυγόμενες επιτροπές, οικονομική, μεταφορών, περιβάλλοντος και βιομηχανίας, να υπάρχει προσωπικό το οποίο θα ασχολείται με αυτό αποκλειστικά για να μπορεί να στηρίξει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μας έχει ζητηθεί βεβαίω τώρα και έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να μειώνουμε το προσωπικό μας αναέτο κατά 1%. 5% μέσα σε 5 χρόνια. Θα πρέπει να, να επιστρέψουμε και 57 μέλη του προσωπικού. Δηλαδή θέσεις οργανογράμματος. Άρα πολλοί που θα, ε, πολλές θέσεις όπου το προσωπικό θα συνταξιοδοτηθεί, θα συνταξιοδοτηθεί δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις καλύψουμε πλέον. Και θα είναι δύσκολο να καλύψουμε αυτά που μόλις εξήγησα μέσω redeployment, κινητικότητας δηλαδή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα εσείς έχετε το λόγο. Ο κύριος Μοκαπρώτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα και τους άλλους που πήραν το λόγο εδώ σήμερα για τόσα μας είπαν όσον αφορά τον προπολογισμό 2016. Από αυτά που άκουσα για τις δαπάνες για το κύριο Κάντ στο Λουξεμβούργο, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε τι λύσεις θα αποφέρουν ε, εξοικονόμηση στο μέλλον. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εμείς δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό. Και αυτά είναι πράγματα λοιπόν που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Επίσης είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το 20% όσον αφορά το διοικητικό κόστος. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πρακτική που ίσως δεν τα καταφέραμε μία φορά τα τελευταία δέκα χρόνια, ε, δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό. Κύριε Γενική Γραμματέα, αναφερθήκατε στους κανόνες, αναφερθήκατε στην περίπτωση των μισθών των βοηθών. Όταν θέλει κάποιος να αυξήσει 100 ευρώ τον μισθό αυτό και όταν είναι κάποιος ο οποίος προηγουμένως είχε υψηλές αμοιβέ, αν δεν τον πληρώσετε αρκετά καλά ε, θα το χάσετε. Οι εμπειρογνώμονες που έρχονται και μας βοηθούν στο έργο μας ως βοηθή. Γι' αυτό λοιπόν πραγματικά θα ήθελα να το δούμε πολύ προσεκτικά αυτό το σύστημα. Και εσείς πιστεύω ότι κληρονομήσατε κάποιους βοηθούς και καταφέρατε να βελτιώσετε το σύστημα αρκετά. Και εσείς διαπιστώσατε ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε μηχανισμούς που να αντιμετωπίσουμε μείωση το μισθών για παράδειγμα ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου δυσλειτουργίας. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι η βελτίωση παρετέρω μπορούμε να επιφέρουμε είναι θετικό. Δεν έχουν καλυφθεί όλα τα αποθεματικά ακόμα πλήρως. Μην ξεχνάμε τι είπε και για το 2013 το ελεκτικό συνέδριο που είπε ότι ο προπολογισμός είναι επικεντρωμένος στο κόστος, τις δαπάνες πολύ περισσότερο από ό,τι στα αποτελέσματα και στα ωφέλη από αυτόν. Ίσως αυτό να μην είναι ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι όλοι εμείς που πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε τη δουλειά για την οποία μας εξέλεξε ο κόσμος, το νομοθετικό έργο δηλαδή, δεν θα πρέπει να ασχολιόμαστε με τα πράγματα τα οποία μας ζητάνε τα μέσα ενημέρωσης να ασχοληθούμε, για παράδειγμα, ή με φούσκες οι οποίες φουσκώνουν, φουσκώνουν, φουσκώνουν. Το έχω πει και άλλη φορά ότι πρέπει να είμαστε εμείς εκείνοι που θα πάρουμε τις πρωτοβουλίες να μειώσουμε το κόστος και να επικεντρωθούμε στο νομοθετικό μας έργο. Ο προπολογισμό δεν πρέπει να αυξάνεται πολύ. Αναφέρθηκα στις μπλε κάρτες, στις τροπολογίες που υποβάλλονται, να έχουν ήδη εγκριθεί Υπάρχουν δηλαδή τρόποι για να κάνουμε παρετέρω εξοικονόμηση, να μην χρησιμοποιούμε τόσο πολύ το χαρτί, να μην τυπώνουμε δηλαδή κείμενα. Για να μην χρειάζεται μεγάλη αύξηση στον προπολογισμό κάθε χρόνο, ο είπε ότι τρέχουσες δαπάνες θα πρέπει να μειωθούν μέχρι 2%. Αυτό το 2% όταν ήταν ο πληθωρισμός 2% ήταν διαφορετικά. Τώρα ο πληθωρισμός θα είναι από ό,τι φαίνεται 1,1 στην Ευρωζώνη. Άρα η κατάσταση είναι διαφορετική με αυτά τα δεδομένα. Συνεπώς, κύριε Γενική Γραμματέα, αν θέλουμε να στηρίξουμε την δίκηση και την διοικητική μας ικανότητα, πρέπει να ακολουθήσουμε την υποχρέωση που αναλάβαμε για μείωση 1% στη δίκηση. Αλλά υπάρχουν και άλλες απαιτήσει για σημείο που χρειάζεται περισσότερο προσωπικό. Οπότε, εδώ πολύ θα θέλαμε να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια αποθέματα. Από τους 6.000 που έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι θα βρούμε. Κάποιος φεύγει, κάποιος ταξιδοτείται, να κάνουμε κάτι δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση για να μην αυξηθεί παρετέρω το προσωπικό μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κάστερ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον που μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψει για τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016, λέει κύριε Γκρέσλερ. Πράγματι, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη δουλειά που κάνουν οι βοηθοί και όχι μόνο ανάμεσα στο αν είναι κάποιος τοπικός ή στο Στρασβούργο ή αλλού, πιο πολύ η διαφορά έχει να κάνει με το αν πρόκειται για διοικητικούς ή όχι. Αυτοί που έχουν την ευθύνη πρέπει να παραμείνουν. Ο κύριος Βίλαντ το είπε ξεκάθαρα. Δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορούμε να πληρώνουμε με τα επιδόματα γραμματείας, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Πράγματι, στη δίκηση μπορούμε να κάνουμε οικονομίες. Ας δούμε τους μισθούς. Οι υπάλληλοι πληρώνονται πολύ περισσότερο από τη βοηθή μας. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να κάνει οικονομίες να δει που μπορεί να κάνει. Δεν μας έχουν εκλέξει για να βοηθήσουμε τη δίκηση να υπάρχει, όχι, αλλά για να κάνουμε τη δίκηση να λειτουργεί ικανοποιητικά και αποτελεσματικά. Συνεπώς χρειάζεται αύξηση. 3.000 ευρώ Στον τομέα του προσωπικού διαπιστώνουμε ότι έχουμε παγώσει τους μισθούς. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν στη συνέχεια οι μισθοί. Αλλά μην το ξεχνάμε ότι έχει υπάρξει αυτό το πάγωμα. Έπειτα πρέπει να δούμε λίγο και πώς αυξάνεται το προσωπικό. Κύριε Γενική Γραμματέα, σας ερωτώ λοιπόν. Μετά τις αυξήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, για πείτε μου, ποιο είναι το οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δει κανεί τα οργανογράμματα, να δει δηλαδή ποιοι είναι επισύμβαση. Να δούμε επίση ποιο είναι ο αριθμό των τοπικών βοηθών. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμό τους νομίζω. Ορισμένοι έχουν 45 τοπικούς βοηθούς. Ωραία θα μου πει ε, και λοιπόν. Ναι, εντάξει, και εγώ θα ήθελα να έχω 45. Στη Γερμανία δεν θα μπορούσα. Αυτή είναι η Ευρώπη. Σε κάποιες χώρες ορισμένοι είναι έτοιμοι να δουλέψουν για το 145ο του επιδόματος. Στη Γερμανία δεν ισχύει αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν πρόκειται να καταφέρουμε να ισοπεδώσουμε τις διαφορές που υπάρχουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Γενική Γραμματέα θέλω αύξηση. Θέλω να δεχτείτε τα 3.000 ευρώ και αν θέλετε να κάνετε εξοικονομήσεις, να τις κάνετε εκεί που μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Γκρέσλερ. Ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ για την εξαιρετικά ποιοτική δουλειά, ως συνήθως δηλαδή που έγινε από πλευράς του Προεδρείου, της Γραμματείας και του εισηγητή μας. Εργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο ο κ. Σεζαραντεπρέ και συνεχίζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπερασπίζεται την αρχή ενός προϋπολογισμού νομίμου, νομότυπου όπου επικρατεί πειθαρχία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει για τα λειτουργικά έξοδα να είμαστε σύνομοι και να επικαιροποιούμε τους κανόνες μας. Πέραν αυτού, τα μεταβλητά έξοδα, οι μεταβλητές δαπάνες, κατά τη γνώμη μας, μπορούν να έχουν ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα ως προς το αποτελεσμά τους. Και γι' αυτό υποστηρίζουμε ε, τη βασική αρχή του προϋπολογισμού, ε, δυνάμει της οποίας ε, θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη οποιαδήποτε αύξηση μεταβλητών δαπανών. Χρειαζόμαστε το ελάχιστο αλλά και το απαραίτητο. Εάν δεν έχουμε τα χρειαζόμενα εδώ στο Κοινοβουλίο, τα, το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι πολίτες. Εάν δεν νομοθετούμε σωστά, αυτό επισύρει ένα κόστος που μετακυλίεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Γι' αυτό θα συμφωνήσω απολύτως με την ανάγκη του να έχουμε τα ελάχιστα που χρειαζόμαστε για το βασικότατο ζήτημα των πράξεων κατά εξουσιοδότηση, παραδείγματος χάρη, ή για, την, για το κοινοβουλευτικό μας έργο. Μην ξεχνούμε, οι 28 κράτη-μέλη μας έχουν εκχωρήσει μετά τις συνθήκες της Λισαβόνας αυξημένες αρμοδιότητες και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε στη θέση ε, πλήρως να ασκούμε αυτές τις νέες αρμοδιότητες. Ταυτόχρονα συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουμε αυτά που χρειαζόμαστε και συγχαίρω και πάλι τον εισηγητή που ε, καταθέτει αυτή τη μετριοβαθή πρόταση γύρω στο 2% είναι επικαιροποιήσεις που χρειάζονται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Υπάρχουν πράγματα όπως το διαδίκτυο, το ασύρματο δίκτυο, προφανή ε, σήμερα πράγματα, αλλά θυμηθείτε τι είχε γίνει από πλευράς κάποιων πολιτικών ομάδων στο παρελθόν. Είχαν διαμαρτυρηθεί και τώρα γυρνάνε και μας λένε δεν είναι αξιόπιστο, δεν υπάρχει κάλυψη ε, παντού. Υπάρχουν πάντοτε εξελίξεις και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Σίγουρα μπορούμε εύκολα να ε, εκμεταλλευτούμε δημαγωγικά τον προϋπολογισμό ε, του, του, του Κοινοβουλίου και δεν θα πρέπει να ξέρουμε δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι μόνο ε, ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει, το 1% και το 99% αντιστοιχεί σε απαιτούμενα κονδύλια για την ίδια τη λειτουργία του, του Κοινοβουλίου. Αυτοί που ορισμένες φορές ε, είναι οι πρώτοι που υπερασπίζονται στα λόγια την αξιοπρεπή εργασία για τους εργαζομένους, την αξιοπρεπή εργασία και τους αξιοπρεπούς μισθούς για τους βοηθούς. Οι ίδιοι αυτοί είναι συνήθως που δεν δίνουν τον αξιοπρεπή μισθό ε, σε αυτούς τους βοηθούς. Πολύ εύκολα γίνεται κάποιος λαϊκιστής ε, και χρησιμοποιεί ως πρόσχημα, ως πρόφαση τον προϋπολογισμό για να ισχυριστούν ότι αυτή η αποζημίωση επιστρέφει στον κορβανά του βουλευτή εάν δεν χρησιμοποιηθεί. Όμως ξέρουμε ότι η διαπιστευμένη βοηθή και ε, πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Και δεν μπορεί κάποιος να ε, συνάψει παραπάνω συμβάσεις από αυτά που προβλέπονται. Και φυσικά για τους ε, τοπικούς βοηθούς αλλά και για τους διαπιστευμένους βοηθούς υπάρχουν όρια ε, ως προς το κονδύλι, το διαθέσιμο κονδύλι. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πειθαρχία, να είμαστε υπεύθυνοι για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν. Έχουμε μια πολύ καλή πρόταση μετά την πολύ καλή ε, συνεργασία που υπήρξε ανάμεσα στην, ε, στο Προεδρείο, στη Γραμματεία, των εισηγητή και τους Σκιώδης εισηγητές και είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε την απαιτούμενη πειθαρχία αφενός στον προπολογισμό αλλά και αφετέρου ε, τα δέοντα κονδύλια τόσο ώστε να μπορέσουμε να ε, επιτελέσουμε το έργο και να υπηρετήσουμε τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριο Σάρβαμα. Ευχαριστώ. Θα είμαι ασφάλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω το Γενικό Γραμματέα να κάνει αυτές τις προτάσεις για την ασφάλεια και θα υποστηρίξω πλήρως αυτή τη γραμμή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει όλοι να το δεχτούμε. Για τους τοπικούς βοηθούς νομίζω ότι Ενδεχομένως να τεθεί και ζήτημα μισθών, όμως κατά τη γνώμη μου περί τίνος πρόκειται. Όταν έχουμε πάνω από τρεις ε, τοπικούς βοηθούς στο κράτος μέλος είναι διαφορετική η κατάσταση. Οτιδήποτε υπερβαίνει τον αριθμό των τριών τοπικών βοηθών στο κράτος μέλος είναι υπερβολικό και ε, πρόκειται για πολιτική αυτοκτονία για το, πολιτικό, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ακριβώς ε, αυτά που τροφοδοτούν τα αντιευρωπαϊκά αισθήματα, τέτοιου είδους πληροφορίες. Ε, οπότε δεν νομίζω ότι είναι και τόσο δύσκολο να αλλάξουμε τους κανόνες. Εγώ προσωπικά έχω ιδέες αν χρειαστεί, αλλά νομίζω μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό μεταγενέστερα. Θα Σα ευχαριστούμε κύριε Σάρμα, ο κύριος Βαλή. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω το Ζεράρ Ντεπρέ, τους ε, αντιπροέδρους, του Γενικό Γραμματέα για τις πληροφορίες ε, που μας παρουσίασαν. Δεν θέλω να φανώ λαϊκιστής, όμως ε, θα ήθελα με πάσα διανοητική ειλικρίνεια να καταθέσω και εγώ τη δική μου επιχειρηματολογία. Ξέρουμε με την χρηματοπιστωτική κρίση ότι έχουν προκύψει σοβαρότατοι περιορισμοί και περικοπές μισθών για τους δημοσίους υπαλλήλους σε χώρες όπως η Ιταλία, περικοπές συντάξεων. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προτού εισηγηθούμε οποιαδήποτε αύξηση να εξετάσουμε με μεγάλη σοβαρότητα και ειλικρίνεια ε, τις προτάσεις. Εγώ συμφωνώ για τον τίτλο, για τον τομέα μάλλον 5 και για την, ε, το ποσοστό που προτείνεται, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η προσαρμογή στον πληθωρισμό και το αν θα η αύξηση θα, είναι, θα κυμαίνεται στο 2 ή στο 3%. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε περισσότερο από τη διαπραγμάτευση ότι υπάρχουν ε, περιτά έξοδα, δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλεια, αυτά που προκύπτουν από τον εσωτερικό κανονισμό βεβαίως είναι αδιαπραγμάτευτα όμως. Ταυτόχρονα δεν θα έπρεπε ε, να αναθεωρήσουμε και τον κανονισμό εφόσον ζητάμε από τις χώρες να προβούν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να τροποποιήσουν ακόμη και το σύνταγμά τους. Γιατί λοιπόν είναι τόσο αδύνατο ε, να τροποποιήσουμε τον ιστορικό κανονισμό του Κοινοβουλίου. Θα έπρεπε και αυτό να είναι δυνατόν. πράξης κατ' εξουσιοδότηση. Όντως ο, ελεγκτικός, ε, ο νέος ελεγκτικός μας ρόλος είναι σημαντικός και πρέπει να αναβαθμιστεί το έργο μας. Όμως ε, ισχυρίζομαι ότι Υπάρχουν γραμμές ε, όπως ε, τα ταμεία των πολιτικών ομάδων, οι αποστολές επιδέχονται τροποποιήσεις για να επαναδιαθέσουμε τα κονδύλια και να αποδείξουμε ταυτόχρονα στους πολίτες, οργισμένους πολίτες, πώς επικρατεί αυστηρότητα, εγκράτεια και πειθαρχία. Νομίζω ότι ε, δεν θα ήμασταν πολύ δημοφιλείς αν ακούγαν τη συζήτησή μας και ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο αύξησης ε, των δαπανών. Πιστεύω ότι θα πρέπει ενδεχομένως να προβούμε σε μια αναθεώρηση ε, των επωνομαζόμενων αναγκαίων δαπανών μέσω τροποποίησης του κανονισμού. Νομίζω ότι για τους βοηθούς 21.000 νομίζω ότι ε, είναι, είναι δυνατόν ε, να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο ε, τροποποίησης και σε αυτό το σημείο των κανόνων. ξέρω ότι αυτά που λέω δεν είναι πολύ δημοφιλή εδώ μέσα, εκτός όμως κοινοβουλίου είναι. Ευχαριστώ κύριο Στάχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, έρχομαι από την Εστονία εγώ, που είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρωζώνης, αλλά εξισορροπεί τον προϋπολογισμό καλά. Γι' αυτό και εγώ και οι πράσινοι συνάδελφοί μου χαίρονται που έχει μια τόσο σόφρονα αντιμετώπιση ο εισηγητής πράγματι πρέπει να είναι παραδειγματική η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτούς τους καιρούς που ζούμε. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είμαστε εκλεγμένοι από το κοινό και άρα η σχέση μας είναι άμεση μαζί του. Αν υπάρξει μεγάλη αύξηση στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου καταλαβαίνετε ότι θα αντιδράσει ο κόσμος. Και είναι λογικό αυτό. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αν θέλουμε ένα συμβασμό ανάμεσα στο 2 και το 3% εγώ θα έλεγα ότι εγώ μάλλον θα ψηφίσω πιο κοντά στο 2%. Πάντως εγώ προσωπικά θα μπορούσα να στηρίξω την αύξηση όσον αφορά τις πληρωμές στους βοηθούς, στους δικούς μου τουλάχιστον. Όλοι ξέρουν ότι άλλοι δίνουν λιγότερα. Οι πράσινοι, γενικά μιλώντας, εντάξει, μπορεί κάποιοι να αποφασίσουν μια διαφορετική στάση, πάντως προς το παρόν προς τα εκεί κατευθυνόμαστε. Τώρα το θέμα των τοπικών βοηθών. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε διστακτικοί στον υπάρχουν διαφορές. Αν υπάρχουν κάποιες ανομαλίες στο θέμα των τοπικών βοηθών, ε, ας τα δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία και το τοπικό εκλογικό σώμα θα ανταποκριθεί ανάλογα στις επόμενες εκλογές. Τώρα όσον αφορά το αίτημα για τον έλεγχο των πρωτοβουλειών και των προτεραιοτήτων όσον αφορά την προηγούμενη θητεία. Και εδώ βάζουμε ένα ερωτηματικό για το Βερολίνο. Όσον αφορά την αντιγραφή Αν αντιγράψουμε λοιπόν τα του Βερολίνου, ίσως μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα πληρώνοντας μια και έξω για να μην έχουμε τόκους. Αλλά θα πρέπει να το ερευνήσουμε. Μήπως επειδή είναι πάρα πολύ χαμηλά τα επιτόκια, δεν είναι αυτό το συμφέρον, αλλά συμφέρει να πληρώνουμε επιτόκια Πρέπει να το ελέγξουμε δηλαδή αυτό. Τέλος, το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό ανάμεσα στο Προεδρείο και την Επιτροπή μας. Και το συμβασμό αυτό να δούμε πώς θα τον μεταφέρουμε προς τα έξω. Γιατί αν πούμε ότι αυξήσαμε 2% τον ε, προπολογισμό μας και ότι σύμφωνα με τα μαθηματικά του Συμβουλίου θα μπορούσαμε να ανέβουμε στα 5%, ε, καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση που δημιουργείται κάθε φορά είναι διαφορετική. Ο κύριος Κολμέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ και τον εισηγητή, αλλά και τους αντιπροέδρους, όπως επίσης και τον Γενικό Γραμματέα. Ανταλλάξαμε απόψεις και θα ήθελα με τη σειρά μου να συνοψίσω λίγο την άποψη της ομάδας μου και τη δικιά μου την άποψη πιο προσωπικά. Να σας πω δηλαδή τι πιστεύω ότι είναι το σημαντικό. Βρισκόμαστε στο κέντρο προσοχής του κοινού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όντως παραδειγματικοί όσον αφορά τις οικονομίες που κάνουμε. Δεν πρέπει να ξεπεράσουμε το 2% στην αύξηση των δαπανών μας. Τα υπόλοιπα θα πετήσουν συζητήσεις και όπως πάντα όταν έχει κανείς αρκετά χρήματα μπαίνει και στον πειρασμό να τα ξοδέψει. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ τα ποσά. Όλοι συμφωνούμε για το ότι πρέπει να κάνουμε κάτι όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφορικής, διότι υπάρχουν και απειλές. Κανείς μας δεν μπορεί να εκτιμήσει επακριβώς τις απειλές αυτές. Μόνο οι ειδικοί μπορούν να το κάνουν. Αλλά διαβάζοντας τις εφημερίδες διαβάζουμε φοβερά σενάρια και θα έπρεπε να είμαστε ε, προετοιμασμένοι. Υπάρχει φυσική μας ε, ασφάλεια και προστασία. Υπάρχει το θέμα της πρόσβασης στα κτίρια αλλά μην καταλήξουμε να έχουμε και ένα πλασεμπό, να μας εξυπηρετεί ιδέα και μόνο, να δούμε πού θα τοποθετήσουμε τα χρήματά μας. Ασφάλεια απόλυτη, έτσι κι δεν υπάρχει. Πρέπει να δεχτούμε μια σχετική ασφάλεια με ποσά που να είναι αποδεκτά. Έτσι κι θέλουμε το κοινοβούλιο να είναι ανοιχτό. Έχουμε ένα σωρό επισκέπτε. Δεν πρέπει να διπλωνόμαστε. Το σημαντικότερο είναι το κόστος προσωπικού για τους βοηθούς. Νομίζω ότι και εδώ πρέπει να δείξουμε θάρρος. Να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις ως Ευρωκοινοβουλίο, διότι πραγματικά δεν κατανοώ πώς είναι δυνατόν κάποιος να απασχολεί δωδεκάδες απασχολουμένους. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Ούτε είναι και η υπόθεση των ξεχωριστών βοηθών, διότι εδώ αμφισβητείται το κύρος του ίδιου του Κοινοβουλίου. Να δώσουμε λοιπόν σε κάποιο εύρος κάποιες κατευθύνσεις πόσο θα είναι το ποσοστό που θα δαπανάτε για διαπιστευμένους βοηθούς και ποιο θα είναι το ποσοστό για τους τοπικούς. Και να ρωτούμε και ποιο είναι το επίπεδο των μισθών στη συγκεκριμένη χώρα. Φαίνεται πως υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που έχουν 43 συνεργάτες. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατον να ε, απασχολήσει ας πούμε στη Γερμανία κάποιος ένα τέτοιο, ποσό, ένα τέτοιο αριθμό ε, συνεργατών. Αυτά πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να υπάρξει και το περιθώριο να μην αυξηθεί μεν το ποσό, αλλά να μπορέσουν να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες, εν πάση περιπτώσει, να προσβληθούν περισσότερα πρόσωπα. Ο κύριος Χριστοφόρου παρακαλώ. Στο κύριε Πρόεδρε, ε, πολύ ορθές οι εισηγήσεις των αγαπητών συναδέρφων. Να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Ντεμπρέ, τον εισηγητή έκθεση, αλλά και τους αντιπροέδρους και τον Γενικό Γραμματέα που βρίσκονται εδώ, για να μας δώσουν έτσι μια εκτενή ενημέρωση του θέματος. Όμως θα υπενθυμίσω δύο-τρία βασικά ζητήματα. Πρώτον, δεν πρέπει να μα διαφεύγει το γεγονό ότι ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μόνο το 2% του συνολικού προπολογισμού αν θέλουμε να κάνουμε πραγματικά νοικοκύρεμα, πιστεύω ότι το νοικοκύρεμα το ξεκινά από το 98% και όχι από το 2%. Έχουμε μεγαλύτερα περιθώρια να κάνουμε νοικοκύρεμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού από το τεράστιο ποσό που διατίθεται για άλλου σκοπού παρά από τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ πιστεύω ότι και αυτό α μην χαρακτηριστεί ή λαϊκιστικό ή αντιλαϊκιστικό, ότι αυτό που απασχολεί τον κόσμο δεν είναι εάν έχει αύξηση ή αυτή τη στιγμή όλο ο κόσμο και η Ευρώπη ασχολείται αν θα έχει αύξηση 2 ή 3% ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που ασχολείται ο κόσμο είναι αν αυτό το κοινοβούλιο είναι αποτελεσματικό. Εάν με το 3% το κοινοβούλιο είναι αποτελεσματικό, σα διαβεβαιώνω ότι θα εξοικονομήσουμε πολύ περισσότερε δαπάνε από ότι πιθανώ με ένα δύο που μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό το κοινοβούλιο. Γνωρίζετε πολύ καλό ότι για να μπορέσουν να αποδώσουν οι υπηρεσίε και να έχουμε ένα σύγχρονο αποτελεσματικό Ευρωκοινοβούλιο, χρειάζονται χρήματα. Και πιστεύω ότι αν αυτά τα χρήματα είναι για παραγωγικό και αποτελεσματικό σκοπό, σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Εάν το δικό μα το κοινοβούλιο δεν είναι αποτελεσματικό και δεν ασκεί το σωστό έλεγχο, χάνονται πάρα πολλά χρήματα. Θα σα μεταφέρω και την εμπειρία τη χώρα μου, όπου ουσιαστικά δεν βρέθηκε σε μνημόνιο γιατί αυξήθηκε ή μειώθηκε ο προπολογισμό 2, 3 ή 5%, αλλά για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπήρχε ένα αποτελεσματικό έλεγχο είτε στι δαπάνε, είτε ακόμα και στα έσοδα που επαρήγονται. Άρα πιστεύω είναι λαθασμένα να επικεντρωθούμε και να θεωρηθεί μείζον θέμα εάν η αύξηση του προπολογισμού θα είναι 2-3%, αλλά πολύ περισσότερο πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, πόσο θα αποδώσουν και πόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και πιστέψτε με και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν επικεντρώνεται στο πόσο εμείς θα αυξήσουμε ή θα μειώσουμε τον προπολογισμό μας αλλά τι έργο θα του προσφέρουμε και τι εικόνα θα δημιουργήσουμε. Και εγώ θα πω ότι με έπεισε ο Γενικό Γραμματέα ότι υπάρχουν ανάγκε και ότι γίνεται σωστή δουλειά προ την κατεύθυνση τη αξιοποίηση των χρημάτων του προπολογισμού. Και πιστεύω ότι εκεί που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα είναι στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των κονδυλίων, όχι μόνο για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και για το υπόλοιπο κομμάτι του ευρωπαϊκού προπολογισμού που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριο Συγκρέσκου, τελευταίος. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Νεγκρέσκου. Θα αναφερθώ στο θέμα των μισθών των βοηθών. Άκουσα διαφορετικές οπτικές γωνίες. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να αναφερθούμε και στο εκλογικό σώμα το οποίο εκπροσωπούμε εδώ. Για τους Ρουμάνους ευρωβουλευτές έχουμε 23 εκατομμύρια στη χώρα μας. ...240.000 χιλιόμετρα. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη, στα 240 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στον πληθυσμό, χρειαζόμαστε πολλούς βοηθούς. Η κριτική που ακούγεται είναι ότι κανείς δεν ξέρει για μας, κανείς δεν ενημερώνεται για το τι κάνουμε εδώ, για το ότι τους εκπροσωπούμε και δουλεύουμε για αυτούς. Άρα το θέμα που τίθεται δεν είναι το κατά πόσο πρέπει να έχουμε περισσότερους ή λιγότερους βοηθούς. Το θέμα που τίθεται είναι ότι πρέπει να έχουμε βοηθούς που να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι τα νούμερα που νοιάζουν. Άκουσα κάποιο συνάδελφο εδώ από τη Γερμανία που έλεγε ότι δεν καταλαβαίνει πώς είναι δυνατόν να μπορεί να έχει κάποιος τόσο πολλούς τοπικούς βοηθούς στη χώρα του. Ε, λοιπόν, Ρουτ απαγορεύει σε μας να πληρώνουμε στη χώρα μας πάνω από χίλια ευρώ για τον ε, μισθό. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη διαφορά, διάκριση μεταξύ των ίδιων των ευρωβουλευτών και μας αναγκάζει να απασχολούμε περισσότερους γιατί το μέγιστο ποσό που μπορούμε να πληρώσουμε ακαθάριστο είναι 1000 ευρώ στο κάθε βοηθό μας. Εγώ είμαι κατά αυτής της διάκρισης, αλλά υπάρχει. Επίσης, αναφερθήκαμε στις δραστηριότητές μας, ημών των Ευρωβουλευτών είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι αμφισβητεί ο κόσμος το ποσό που δαπανάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που αμφισβητούν είναι τις δραστηριότητές μας, κατά πόσο αυτές είναι χρήσιμες για τους πολίτες. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα όμως πρέπει να έχουμε πολιτικό προσωπικό. Και εδώ στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο, αλλά και πολιτικό προσωπικό με ψηλά προσόντα, πολύ καλά προετοιμασμένο και στις χώρες μας. Οπότε, συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τουλάχιστον έναν ή δύο βοηθούς εδώ, αλλά δεν μπορεί κανείς να μας υποχρεώσει να έχουμε μόνο δύο βοηθούς στις χώρες μας, γιατί τους πολίτες από τις χώρες μας εκπροσωπούμε εδώ. Μην το ξεχνάμε εξάλλου ότι στα συντάγματά μας υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Σας είπα, για 170 εκατομμύρια και 240 ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα δεν μπορούμε να εκπροσωπηθούμε από δύο βοηθούς. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους αντιπροέδρους και στο Γενικό Γραμματέα βέβαια και θα ζητήσω και από τον εισηγητή, τον Ζεράρ Πρέ, να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τις παρεμβάσεις τους. Προηγουμένως όμως εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, οι παρατηρήσεις που ακούσαμε σήμερα μαρτυρούν το εξής. Αποφασίζοντας να είμαστε εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, κάναμε μια δύσκολη επιλογή και άχαρη. Ο προϋπολογισμός δίνει την σκληρή πραγματικότητα. Αυτή μας εμφανίζει. Αυτό το οποίο με εκπλήσει είναι ότι έχουν ληφθεί πολύ σημαντικές αποφάσεις πριν από τρία χρόνια. Αποφάσεις βάσει των οποίων αποφασίσαμε ότι τα έξοδα προσωπικού πρέπει να μειώνονται 1% ετησίως ότι κατά συνέπεια το προσωπικό αποφάσισε να περάσει από τις 35-40 ώρες την εβδομάδα, από 37-40, και η σύνταξη από τα 62 που ήταν έφτασε στα 65-67. Πρόκειται δηλαδή για πολύ σημαντικές και σοβαρές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει και αλλαγές στο καταστατικό του προσωπικού. Και διαπιστώνουμε επίσης ότι παρά τις αλλαγές αυτές δεν έχουμε καταφέρει τα αποτελέσματα που θέλαμε. Φανταστείτε και να μην τις είχαμε κάνει. Είναι το πρόβλημα το καταστατικό. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής που μας το επιθυμίζει συνήθως, κάποιες χώρες σήμερα είναι αναγκασμένες να κάνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να αποτελεί το φυτόριο των ε, διευθυντικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς φυσικά να πλήτεται η ικανότητά του να παράγει έργο με καλές επιδόσεις. Θέλω επίσης να εκφράσω την επιθυμία να μπορούμε, αν μη τι άλλο μεσοπρόθεσμα, να βλέπουμε ποια θα είναι η κατάσταση. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών συμμετέχω στο διοικητικό Συμβούλιο του οίκου Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Και οφείλω εδώ να σας πω ότι δεν είναι πολύ εύκολο να προβλέψουμε τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να μπορούμε να στηριχτούμε σε δημοσιονομικές προβλέψεις τουλάχιστον για μία πενταετία όταν πρόκειται να κάνουμε επενδύσεις και θα ήθελα να έχουμε αρκετά συγκεκριμένη εικόνα για τις επενδύσεις αυτές και για το πώς θα χρηματοδοτηθούν. Όσοι συμμετέχουν στο Διοικητικό αυτό Συμβούλιο δυσκολεύονται να δεχτούν ότι θα πρέπει να ελέγχουμε αυτούς που μπαίνουν στο νίκο αυτό της ευρωπαϊκής ιστορίας γιατί λένε είναι κάτι σαν μουσείο πρέπει να είναι ανοιχτό. Εκφράσαμε επίσης την επιθυμία να μπορούμε τουλάχιστον σε πέντε χρόνια να έχουμε προβλέψεις επενδύσεων. Σήμερα μπορεί να δεχτούμε κάποια εξέλιξη των ε, τρέχουσών ε, δαπανών, των λειτουργικών δαπανών δηλαδή. Πρέπει όμως να είμαστε σε θέση και αύριο και μεθαύριο να μπορούμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση όταν θα μας έρθουν νέες δαπάνες. Εγώ κατάλαβα ότι το συνταξιδοτικό μας σύστημα δεν ε, έχει εξασφαλισμένη την χρηματοδότησή του και ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να προσθέσουμε εκεί κονδύλια τα οποία θα προσθεθούν στις άλλες τρέχουσες δαπάνες που έχουμε ήδη προβλέψει. Οπότε η επιθυμία που εκφράζω εγώ είναι να υπάρχει προβλεψιμότητα στον προϋπολογισμό τα επόμενα χρόνια. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι πήραν το λόγο εδώ και ιδιαίτερα τον εισηγητή μας, τους αντιπροέδρους μας και τον γενικό μας γραμματέα. Οπότε, σας παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριο Σασόλη πρώτα. Ευχαριστώ. για την ε, συζήτηση που κάνουμε. Ε, ό,τι ακούσαμε νομίζω σχετίζεται με τρία βασικότατα ζητήματα του προϋπολογισμού. Ε, εργαστήκαμε σκληρά για να καταλήξουμε στις κατευθυντήριες γραμμές. Όλοι δικεύεστε σε δημοσιονομικά ζητήματα και ξέρετε ότι άλλο η δουλειά που κάνουμε εδώ και άλλο αυτά που θα διαβάσουμε στον τύπο και θα ακούσουμε από την κοινή γνώμη. Νομίζω ότι με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή σας μπορούμε να πούμε πως ε, αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό που χρειαζόμαστε για το κοινοβουλευτικό μας έργο. Όταν ε, μιλούμε για τους βοηθούς και ξέρω ότι αυτό το, ζήτημα θα απασχολήσει περισσότερο τον τύπο για πολιτικούς λόγους, δεν ε, ζητούμε αύξηση της βουλευτικής αποζημίωσης των μισθών μας. Ζητούμε μόνο αυτά που μας επιτρέπουν να επιτελέσουμε το έργο μας. Οι βουλευτές θα κληθούν να πάρουν την απόφαση και ήθελα να σας πω κυρία Γκρέσλε πως ε, το ζήτημα όπως το θέσατε Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και σε θέση να εξηγήσουμε στους πολίτες περί τίνος πρόκειται. Δεν πρόκειται για επίδομα, πρόκειται για παρασχεδίες υπηρεσίες, για συμβάσεις εργασίας. Ε, είναι και παιδαγωγικό το έργο μας, θα πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα ε, τι, τι επιδιώκουμε. Οι πολιτικές ομάδες ε, θα πάρουν τις αποφάσεις τους, όμως ξεκάθαρα τα στοιχεία είναι αυτά που εκθέσατε και εσείς και ο εισηγητής. Για τις αυξήσεις στον προϋπολογισμό έχει αποχωρήσει το μεταξύ ο κύριος Τάραντ, αλλά δεν θα ήθελε να δημιουργηθεί σύγχυση. Ο κύριος Ντεπρέ μας εξήγησε με σαφήνεια ότι ε, αυτό στο οποίο αποσκοπούμε είναι 2% αύξηση για τα λειτουργικά έξοδα. Είναι η μισθή, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή, οι συντάξεις. Δεν έχουμε άλλη επιλογή φέτος. Χρειάζεται επίσης και ελπίζουμε να είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα για να μην ε, ανακύψει και πάλι η ανάγκη σε 3-4 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν το έργο κατοχύρωση της ασφάλειάς μας. Μία φορά κάθε 10 ή 20 χρόνια θα χρειάζεται παρέμβαση. Όχι κάθε δύο χρόνια. Είναι όλα τα κτίρια μας ευπρόσβλητα. Είμαστε εκτεθειμένοι σε κινδύνους. Όλες οι υποδομές που έχουμε είναι εκτεθειμένες το σύστημα πληροφορικής, τα κτίρια μας. Πρέπει να επενδύσουμε. Χρειαζόμαστε κονδύλια για να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια, για να θωρακιστούμε. Ο κύριος Ντεπρέ έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να κάνουμε σαφέστα διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις δύο βασικές γραμμές ε, του προϋπολογισμού, τα λειτουργικά έξοδα και τα επιπρόσθετα έξοδα, τα έκτακτα έξοδα. Ξέρετε, ένα καλό κοινοβούλιο εξορθολογίζει τις υπηρεσίες, δεν περικόπτει μισθούς. Με τον αντιπρόεδρο Βίλαντ και ολόκληρο το Προεδρείο συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κακές συνήθειες στο Κοινοβούλιο. Ο τομέας της εστίασης, παραδείγματο χάρη, στο Κοινοβούλιο ε, ανατίθεται εδώ και 25 χρόνια σε μία εταιρεία, σε, στους τρεις χώρους εργασίας. Συγγνώμη, είναι ε, λογικό, είναι καλή πολιτική. Ζητούμε λοιπόν την υποβολή προσφορών, τη διεξαγωγή διαγωνισμών, προσφορές από όλα τα κράτη-μέλη, όπως ακριβώς γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κάνουμε λοιπόν το διαγωνισμό, διαγωνισμούς μάλλον, για την αναδιάρθρωση αυτή που χρειάζεται. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η διαδικασία και ξέρετε ότι μέχρι στιγμής ε, στη διαδικασία του ε, διαγωνισμού δεν θα αναλαμβάνουμε εμείς πλέον τους κινδύνους για την εταιρεία, τον ανάδοχο, την ανάδοχη εταιρεία. Ε, Ξεκονομούμε έτσι ένα εκατομμύριο από τα, τις δαπάνες. 1,6. Χρειάζεται η, προσαρμο... η αναπροσαρμογή διότι είναι και διαφορετικές ε, οι αγορές εργασίας ε, ε, όταν μιλάμε για τους βοηθούς. Είναι διαφορετικές οι συμβάσεις ανάλογα με τη χώρα, την Πολωνία, τη Γερμανία, την Ιταλία. Είναι διαφορετικό το κόστος και οι 20, 25, 22, 23 θα πρέπει να ισοδυναμούν με το ίδιο πράγμα για όλους τους 750 βουλευτές των 28 διαφορετικών κρατών μελών. Δίκιο έχει η κυρία Γκρέσλε όταν ζητάει την προσαρμογή αυτή. Όμω οι πολιτικές ομάδες θα το αποφασίσουν γιατί χρειάζεται πρώτερη συνένεση των βουλευτών. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σα και για τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε Αντιπρόεδρε Σασόλου και τώρα ο Αντιπρόεδρος Βίλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε όλη αυτή τη συζήτηση ας αποφύγουμε να επιτρέψουμε να δημιουργηθεί εντύπωση σαν δίθεν οι βουλευτέ να είναι ενάντια στη διοίκηση, η διοίκηση ενάντια στι πολιτικέ ομάδες και το καθεξής. Εν τέλει, όποιο και να φταίει, όπω και στο ποδόσφαιρο, η ομάδα χάνει ολόκληρη. Ορισμένα πράγματα μπορεί να ήταν σωστά και δημοφιλή. Κάποια στιγμή έρχεται όμω που είναι περιτά. Συζητούμε τώρα αν θα προβούμε σε προμήθειες συσκευών που πριν από τρία χρόνια δεν ξέραμε καν αν υπάρχουν, ότι υπάρχουν δηλαδή. Το ίδιο. Με το χαρτί, εξοικονόμηση χαρτιού, διότι γίνονται τα έγγραφα ηλεκτρονικά. Πρέπει να μείνουμε λοιπόν να παρακολουθούμε την εξέλιξη των καιρών. Όπως είπα, όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε. Ούτε είναι και τόσο άσχημο το Ευρωκοινοβούλιο. Για πολλά χρόνια βάλαμε γύρους μηδέν, μηδενικής αύξησης, ιδίως για το επίδομα της γραμματείας. Μάλιστα καμιά φορά ξεπεράσαμε και τους εαυτούς μας στις περικοπές. Δεν λέω ότι έγιναν για λαϊκίστικους λόγους, αλλά έγιναν μερικά πράγματα. Και δεν έχουμε δει ούτε έναν που να ήρθε και να μας είπε «Α, ξέρετε, με επενούν στη χώρα μου, διότι δαπανώ λιγότερα». Δεν ξέρω ούτε έναν βουλευτή που να έλαβε έστω και μία ψήφο παραπάνω επειδή έκανε εξοικονομήσεις εδώ. Ίσως μάλιστα να είναι και το αντίθετο διότι τώρα φτάνουμε σιγά σιγά στα όρια του εφικτού. Και γι' αυτό μας θεωρούν όλο και περισσότερο σαν ανεπαρκείς. Πρέπει τώρα να έρθουμε στο ύψος όμως της Ευρώπης της ε, συνθήκης της Λισαβόνας και ιδίως για το θέμα αυτό των πολιτικών ομάδων και της διοίκησης. Πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση αυτή γιατί υπάρχουν και εξισορροπητικά αποτελέσματα στη δράση μεταξύ διοίκησης και ευρωβουλευτών. Και στους συνεργάτες πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα. Βεβαίως τα νούμερα δεν είναι πάντα συγκρίσιμα. Θα σας πω ένα πράγμα όμως. Το κόστος του κοινοβουλευτικού συστήματος στις ΗΠΑ κοστίζει σε κάθε ε, ε, Αμερικανό φορολογούμενο περίπου 5 ευρώ το χρόνο. Το κόστος του κοινοβουλίου εδώ είναι περίπου 3 ευρώ το χρόνο για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Παρόλο που, και δεν θέλω να ξεκινήσουμε συζήτηση τώρα, πρέπει να δεχτεί αυτό, παρόλο που εμείς στις αποσκευές μας έχουμε και τις τρεις έδρες εργασίας και τη μετάφραση και τη διερμηνία δηλαδή συνθήκες πλαίσια της εργασίας που δεν έχουν οι Αμερικανοί, όπου εμείς δεν μπορούμε να τις επηρεάσουμε, τρεις έδρες εργασίας για παράδειγμα, και όμως επηρεάζουν βαθιά τη δουλειά μας. Αν δεν τα είχαμε όλα αυτά, τα οποία δεν έχουν οι Αμερικανοί, θα είμαστε στα 2 ευρώ επιβάρυνση του κάθε Ευρωπαίου πολίτη το χρόνο, όταν είναι 5 για τους Αμερικανούς. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε και κάποια αυτοπεποίθηση να προσεγγίζουμε τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Εσείς κύριε Γενική Γραμματεύ, στο χρονοδιάγραμμα έχουμε προβλέψει μια προ-συνδιαλλαγή συνδιαλλαγή μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Προεδρείου για τις 24 Τρίτου και μου λένε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αυτή η ημερομηνία. Μπορείτε λοιπόν να μας γνωρίσετε το συντομότερο δυνατόν ποια θα είναι η ημερομηνία αυτής της φάσης προσυνδιαλλαγής. Και η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών έχει οριστεί για τις 19 Τρίτου Μαρτίου. Δηλαδή. Ο Γενικός Γραμματέας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα, ασφαλώς ακούστηκαν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Αν μπορώ να βγάλω ένα κοινό παρονομαστή, νομίζω μπορώ να πω ότι οι θέσεις όσων εκφράστηκαν δεν απέχουν τόσο πολύ. Υπάρχουν κάποια δύσκολα θέματα που πρέπει να επιληθούν, αλλά στο σύνολο νομίζω μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξο. Ότι δηλαδή τα θέματα αυτά όπου δεν έχουν προσεγγίσει απόλυτα ακόμα θα μπορέσουν να λυθούν. Θα έλθω κυρίως στα πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Ο κ. Μάνκα έθιξε το θέμα του πληθωρισμού, δηλαδή ποιο ρυθμό πληθωρισμού πρέπει να βάλουμε σαν βάση για τις σταθερές δαπάνες του Κοινοβουλίου, δηλαδή αυτές όπου ανταποκρίνονται στις απόλυτες υποχρεώσεις που έχει το Κοινοβούλιο. Αυτό φτάνει στο 2,2%. Δηλαδή αποζημιώσεις βουλευτών, κάποιες συμβάσεις, αμοιβέ. Αυτή, αυτός είναι ο ρυθμός αύξησης από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε για τον καθορισμό του προπολογισμού. κυρία Γκρέσλε ρώτησε πού μπορεί να δει κανεί την αύξηση του προσωπικού στο οργανόγραμμα, το οποίο προσαρτάται στον προπολογισμό. Και αν υπάρχουν βέβαια επιμέρους ερωτήσεις, ευχαριστώ να τις απαντήσω. Ο κύριος Φερνάντες αφενός μας είναι χάρη για την πρόταση και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και νομίζω ότι δικαίω τόνισε ότι το πιο δαπανηρό, το πιο ακριβό πράγμα είναι η κακή νομοθετική εργασία. Αυτό θα έχει το μεγαλύτερο κόστο, δηλαδή αν το έπρατε το Κοινοβούλιο. Και ότι ακόμα δεν έχουμε καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας, δηλαδή τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας. Εδώ, σε συνεργασία με τον εισηγητή, θα κάνουμε κάποιες προτάσεις για να ενισχύσουμε τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου. Ο κ. Σαββά μίλησε για την ασφάλεια, τα μέτρα τα στηρίζει, και θεωρεί ότι πρέπει να θέσουμε και το θέμα και εμείς του αριθμού των ντόπιων συνεργατών. Ο κ. Βάλλη είπε ότι τα θέματα αυτά δεν μπορούν να μπουν όλα στο καταστατικό. Αυτό το συζητήσαμε ήδη και πέρσι. Ήδη ο Πρόεδρος σας ανέφερε ορισμένα, ορισμένα από τα μέτρα. Την αύξηση δηλαδή της εβδομάδας εργασίας από 40 σε 42 ώρες την αύξηση του συνταξιοδοτικού ορίου ηλικία βαθμιδών μέχρι τα 66 έτη της ηλικία Κάποια μέτρα δεν αναφέρθηκαν, είναι σημαντικά όμως και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις. Βέβαια εξαρτάται και πώ θα εφαρμοστεί, διότι η σταδιοδρομία φτάνει μέχρι τον διοικητικό βαθμό 12, εκτός αν κανείς έχει ε, υψηλότερε διοικητικέ ευθύνε, κάτι στο ένα επίπεδο δηλαδή στο οποίο οι περισσότεροι υπάλληλοι δεν φτάνουν. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν τέτοιε ιδιαίτερε διοικητικέ ευθύνε, φτάνουν μέχρι τον 12ο βαθμό. Είχαμε ένα σύστημα όπου όλοι μέχρι τώρα προήγονται αυτομάτω μέχρι τον βαθμό 13 ή και 14. Αυτά είναι βεβαίω και ιδιαίτερα. Οι βαθμοί αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλά αμοιβόμενοι και αυτό έχει επιπτώσει και στην σύνταξη. Όμω αυτή η αυτόματη προαγωγή τέλειωσε. Οι επιπτώσεις στους χαμηλότερους βαθμούς είναι βέβαια πολύ περιορισμένοι, αλλά το συσσωρευμένο αποτέλεσμα μέσα από την πάροδο των ετών και στις συντάξεις θα είναι σημαντικό, ώστε με το μέτρο αυτό έχουμε βάλει μια ισχυρή τροχοπέδη στο κόστος. Βεβαίως εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο συνεπώς. Οφείλω να πω ότι έως τώρα, μέχρι σήμερα, Κανένας δεν έχει προαχθεί σε ιδιότητα συμβούλου που σημαίνει ότι από τον 12ο βαθμό θα περάσει στον 13ο και στον 14ο. Άρα μέχρι τώρα η εφαρμογή του μέτρου είναι απόλυτα συνεπής και το συνδέουμε μοναχά με την ανάληψη των καθηγόντων του τμήματάρχου, άρα ιδιαίτερων δικαιωτικών ευθυνών. πάντως με τρόπο που να μην αρθεί πάλι αυτό το τροχοπηδητικό αποτέλεσμα. Αυτό θα είναι και το μέτρο που στο καταστατικό θα έχει και τις μεγαλύτερες επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. Ο κ. Τάραντ επίσης αναφέρθηκε στο Παρλαμεντάριουμ. Την συζήτηση αυτή την έχουμε κάνει για το μέγα το κοινοβουλευτάριον αν επιτρέπετε ο νεολογισμός. Έχουμε 350.000 επισκέπτες και έτσι έχουμε φτάσει να γίνουμε η δεύτερη ή τρίτη ατραξιόν στις Βρυξέλλες. Έχουμε φτάσει άλλωστε και στο όριο αντοχής από άποψη αριθμού επισκεπτών. Μπορεί λοιπόν να είναι σημαντικό εργαλείο και σε ορισμένε χώρες μέλη και κατά τη γνώμη μου όχι και ιδιαίτερα δαπανηρό. Αυτό θα το δούμε βεβαίως. Χρειαζόμαστε ασφαλώς πάρα πολύ ελκυστικούς τόπους όπου να ιδρυθούν αυτά. Βεβαίως η λεωφόρος υπότα φιλήρας στο Βερολίνο είναι ένας τέτοιος τόπος. Είναι περίφημη Unter den Linden. Άλλοι βουλευτές μίλησαν μετά, είπαν ότι έχει καλός για τους ε, βοηθούς όμως είπαν ότι ίσως είναι δυνατόν να υπάρξει και ένα συγκεκριμένο επίπεδο αμοιβών για τους διαπιστευμένους βοηθούς. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσει το Προεδρείο. Ο κύριος Χριστοφόρου με τη σειρά του είπε ότι είναι σημαντικό τα χρήματα που έχουμε να δαπανώνται και με σωστό τρόπο, λογικά και επί της ουσίας και βεβαίως και με ορθό τρόπο και στην απαλλαγή 2013 είχαμε βέβαια την κατάσταση ότι δεν υπήρξε κριτική από πλευρά ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτό βέβαια μπορεί να αλλάξει. Αλλά για την ώρα νομίζω έχουμε επαρκή εχέγγυα ότι αυτοί οι επαγγελματίες ελεγκτές έχουν καταλήξει βέβαια σε θετικό συμπέρασμα. Ο κ. Νεγκρέσκου τόνισε και πάλι την κατάσταση των Ρουμάνων Ευρωβουλευτών και επίσης το γεγονός ότι η ισχύουσα ρύθμιση για το ανώτατο επίπεδο για τους ντόπιου βοηθούς είναι πολύ αυστηρό δηλαδή κάτω από 1000 ευρώ ε, ακαθάριστα, εγώ συμφωνώ. Τέθηκε το θέμα και στο Προεδρείο, δηλαδή με τα προσόντα όπου απαιτούνται για έναν κοινοβουλευτικό βοηθό, νομίζω το όριο αυτό οδηγεί σε διακρίσεις απέναντι σε ευρωβουλευτές ορισμένων χωρών μελών. Γι' αυτό και θα επανεξεταστεί, οφείλεται να επανεξεταστεί το θέμα και στο μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πιο ευέλικτο τρόπο. Ο πρόεδρος, κ. Αρτουή, έθεσε ορισμένες ερωτήσεις για τον βαθμό άντε 12, μίλησα ήδη, είπα ότι θα σημάνει και μια τροχοπέδη στο κόστος και βεβαίω στο μέλλον όλο και περισσότεροι υπάλληλοι θα ε, θίγονται από το μέτρο αυτό, δηλαδή θα ε, επηρεάζονται από το μέτρο αυτό για τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Είπα, ο ετήσιος προϋπολογισμός έχει συμφωνηθεί με την Επιτροπή Προϋπολογισμών στα επίπεδα του 2011 έως 2012. Θα διατηρηθεί οι δαπάνες αυτές, άλλωστε δεν είναι επιπρόσθετες δαπάνες, εφόσον όλες οι οργανικές θέσεις του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας έχουν ληφθεί από άλλες θέσεις δεν έχουμε δηλαδή προσλάβει νέους υπαλληλούς που θα σήμαιναν πρόσθετες δαπάνες. Τους έχουμε πάρει από άλλες υπηρεσίες για να τους θέσουμε στη διάθεση του οίκου της ευρωπαϊκής ιστορίας. Άρα οι αιτήσει δαπάνες δεν είναι επιπρόσθετες. Και μάλιστα υπάρχει και μια τάση μάλλον υπερτίμησής τους παρά υποτίμησής τους. Για, την μακροπρόθεσμο, για τον μακροπρόθεσμο υπολογισμό των δαπανών θα χρειαστεί να, δούμε τι γίνεται και στον τομέα των ακινήτων. Γι' αυτό το Προεδρείο θα κληθεί να ασχοληθεί με την μεσοπρόθεσμη πολιτική ακινήτων. Υπάρχει η ομάδα εργασία ακινήτων με την Προεδρία του Αντιπροέδρου Βίλαντ που έχει καταθέσει σχετική πρόταση η οποία θα μας επιτρέψει να δώσουμε και πλέον συγκεκριμένες πληροφορίες για τις αναμενόμενες εξελίξεις του κόστους για τα επόμενα έτη. Για τις συντάξεις, για τις συντάξεις έχουμε ορισμένες απαλλαγές. Η Κομισιόν περιέλαβε στον προπολογισμό και τη συντάξη των βουλευτών, όμως εξακολουθεί να είναι μετέωρο το θέμα του πρώην εθελοντικού συνταξιδοτικού ταμείου των Ευρωβουλευτών. Εκεί πρέπει να βρεθεί κάποια λύση στον προπολογισμό. Σας ευχαριστώ και για την Έχω συνεννοηθεί με τον εισηγητή για μια πρώτη συνάντηση την Τετάρτη και με του αντιπροέδρους θα καταστρώσουμε το, το χρονοδιάγραμμα για το πότε θα διεξαχθούν ποιες συνεδριάσεις. Θα ήθελα να ακούσουμε τον ε, εισηγητή μας. Ε, μπορείτε να αντλήσετε συμπεράσματα από αυτή τη διαφωτιστική και ομολογουμένως πλουσιότατη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, εφόσον ε, ο Γενικός Γραμματέας ε, μας έκανε την τιμή να απαντήσει στα περισσότερα από τα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι. Τρία είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγω εγώ μετά τη συζήτησή μας. Πρώτον, δεν νομίζω πως τη συζήτηση που θα γίνει ανάμεσα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και ε, το Προεδρείο να ε, επιμείνουμε μόνο σε αυτά τα κονδύλια που χρειάζονται ούτως ώστε να εκπληρώσει ε, το Κοινοβούλιο της υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας και των υπολείπων. Εγώ νομίζω ότι για τη δεύτερη κατηγορία ενδεχομένως να προκύψουν τα περισσότερα προβλήματα. Δεύτερον, Νομίζω ότι υπάρχει συνέντευξη σε σχέση με τι βασικέ κατευθυντήριε γραμμέ που έχω εισηγηθεί εγώ, ίσω με κάποιε μικροπροσαρμογέ. Προτού όμω ξεκινήσω τι διαπραγματεύσει, θα ήθελα να γνωρίζω ε, ακριβώ ποια είναι η θέση μα, διότι με το που οριστεί η ημερομηνία πρόεδρε θα αρχίσουν διαπραγματεύσει και θα ήθελα να ξέρω εάν για τους βασικούς προσανατολισμούς και για τους, τα ποσοστά και τα νούμερα που προτείνω, έχω την συγκατάθεση της Επιτροπής μας. Εξηγούμε. Είναι πολύ απλό. Σήμερα έχουμε θέσει στόχους και προτεραιότητες. Δεν είπα όμως τίποτα εγώ προσωπικά για την ε, εξοικονόμηση πόρων. Δηλαδή ούτε ένα μέτρο μείωσης δεν πρότεινα. Ό,τι ακούσαμε σήμερα επισύρει αύξηση στον ε, προϋπολογισμό. Θέλω λοιπόν να το ξεκαθαρίσω. Εάν εσείς μου δώσετε τη συγκατάθεσή σας ότι δεν θα ξεπεράσουμε το 1,9% για τα τρέχοντα έξοδα ενώ η πρόταση του Γενικού Γραμματέα κυμαίνεται στο 3,9% θα, θα πρέπει να εκπονοήσουμε 21 εκατομμύρια. Αυτόματα. Είναι μαθηματικό. Μπορώ από τα 21 εκατομμύρια να αφαιρέσω κάποια πράγματα που έχει προϋπολογίσει ως τρέχοντα έξοδα ο Γενικός Γραμματέας στην πρότασή του, την ασφάλεια των εκτηρίων, την κυβερνοασφάλεια κτλ. 7 εκατομμύρια είναι αυτά. Υπολείπονται 15 εκατομμύρια εάν ε, βασιστούμε στα ποσά που προτείνω εγώ. 15 εκατομμύρια πρέπει να εξοικονομηθούν και ε, χωρίς συναισθηματισμούς θα ήθελα να σας πω ότι Ακόμη και αν δεν θέλετε να αυξήσετε το, την αποζημίωση, γιατί ξέρω ότι ο Γενικός Γραμματέας το έχει προϋπολογίσει αυτό. Αν θέλουμε να, να υπερβούμε, αυτές τις προβλέψεις, ε, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε επιπρόσθετο, αυτό εννοώ, θα πρέπει να προσθεθεί στα 15 εκατομμύρια που πρέπει ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως συγγνώμη, να εξοικονομήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε συμφωνία για αυτό το κεντρικότατο ζήτημα. Το ρυθμό αύξηση, το πόσο αύξηση ε, της ε, γραμματιακής υποστήριξης δηλαδή από το 1,9% και μετά, ό,τι προσθέσετε θα πρέπει να το κόψετε από αλλού. Θαύματα δεν γίνονται. Θα πρέπει λοιπόν, προτού ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με το Προεδρείο, να προτείνουμε και τα μέτρα μείωση ε, των δαπανών για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στο πλαίσιο που εξέδεσα σήμερα. Ξαναλέω, όσο αυξάνεται η αποζημίωση, τόσε περισσότερες θέσεις θα πρέπει να συμπιέσουμε και να ε, περικόψουμε. Είναι ε, μαθηματικά αναπόφευκτο και θα πρέπει να το ξέρετε. Σας είπα ότι ε, από τα 21 εκατομμύρια βάζουμε τα 7 στον έκτατο προϋπολογισμό, υπολείπεται ένα ποσό των 15 εκατομμυρίων που πρέπει οπωσδήποτε να εξοικονομηθεί. Ας επομιστούν όλες τις ευθύνες τους λοιπόν. Δεν αμφισβητώ, προσέξτε, δεν αμφισβητώ ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ακριβώς όπως λέμε στο διεθνές εμπόριο ε, τους ε, θεμητούς όρους για τις συναλλαγές μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Έτσι, λίγη συζήτηση για το ε, σχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2016. Θα επανέλθουμε στη συνάντηση των συντονιστών που θα λάβει η χώρα μόλις λήξει η συνεδρίαση της Επιτροπής στο θέμα της διαπραγματευτικής εντολής για την προσυνδιαλλαγή με το Προεδρείο θα πρέπει να δούμε την ημερομηνία διότι η ενδεικτική ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει προβλεφθεί για την 16η Απριλίου. Στις 27 Απριλίου προβλέπεται η έγκριση του σχεδίου των προκατακτικών δηλαδή προβλέψεων και 27-28 Απριλίου τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Ολομέλεια τέλη Μαΐου. Είναι πάρα πολύ στενό το χρονικό περιθώριο που έχουμε. Στις 16 Απριλίου θα πρέπει να αποφανθεί η Επιτροπή Προϋπολογισμών και άρα θα ήθελα η προσυνδιαλλαγή να ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, ούτω ώστε να έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για να επιτύχουμε σύγκληση στο μέτρο που θα είναι μεγάλη απόκληση των αρχικών απόψεων. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους ε, για την παρουσία τους, για τις δηλώσεις που έκαναν ούτω ώστε να μας διαφωτίσουν στα πλαίσια της προετοιμασίας της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Σας ευχαριστούμε. Monsieur le Président. Bien, nous allons aborder maintenant le projet de budget rectificatif numéro 2 pour 2015. Περνάμε στο διευθυντικό προπολογισμό για το 2015 που έχει να κάνει με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έκθεση Holbridge και Τόμα. Η κυρία Κόντρα Θαμπάλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, είμαστε πολύ πίσω στην ημερήσια διάταξη, οπότε δύο λόγια θα πω μόνο. Πρόκειται για την τροποποίηση του ε, κανονισμού όσον αφορά το 2015 του πολιτισμού δημοσιονομικού πλησίου για το 2015 έχει να κάνει και με το Ταμείο Συνοχής. Υπάρχει μία παράγραφο στην πρόταση αυτή όπου λέμε ότι συμφωνούμε απόλυτα ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί να περάσει στο 2015. Όμως, δείχνουμε και έτσι ξεκινάμε, την ανησυχία μας που είναι όλο και μεγαλύτερη κάθε χρόνο για την καθυστέρηση στην, ε, στις πληρωμές, στην εκτέλεση του προπολογισμού κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε η Γενική Συγκήτρια. Ποιος θέλει το λόγο? Κανείς? Παρακαλώ. Ο κύριος Μουρισάν. Ευχαριστώ εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας. Φυσικά και χαιρόμαστε για την απόφαση αυτή της Επιτροπής να μεταφέρει τις πιστώσεις και συμμερίζομαι και τις ανησυχίες της εισηγήτριας όσον αφορά τον αντίκτυπο τελικά που έχει κατάσταση στις πληρωμές. Έχω όμως και μια δεύτερη ανησυχία που έχει να κάνει με τις υποχρώσεις. Δεδομένου ότι καθυστερεί η έγκριση των προγραμμάτων από πολλές χώρες, οι υποχρεώσεις για το 2015 διπλασιάζονται. Βλέπω λοιπόν έναν μεγάλο κίνδυνο η Επιτροπή θα έπρεπε να είναι ευέλικτη έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τις υποχρώσεις. Ευχαριστούμε, κύριο Χόλμπριχτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να υπογραμμίσω ότι εδώ έχουμε δύο παράλληλες διαδικασίες και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, το είπατε και εσείς στην αρχή. Η μία διαδικασία είναι οι αλλαγή στον προπολογισμό του 2015 και εκ παραλίλου έχουμε την αναθεώρηση της κυρίας Τομά. Επίσημα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στην ουσία όμως είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Και γιατί. Γιατί πρόκειται για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει εκεί η δυνατότητα μεταφοράς των υποχρεώσεων εφόσον τα προγράμματα δεν είναι έτοιμα. Και υπάρχουν τα προγράμματα που είναι έτοιμα, εκείνα τα οποία είναι σχεδόν έτοιμα, που αυτόματα πάνε στο 15 και εκείνα που δεν είναι έτοιμα. Και αν δεν την κάνουμε την μεταφορά, το πρόβλημα δεν είναι μόνο για το 15, είναι και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γιατί ο κανόνα του νησιν 3 εδώ παίζει σημαντικό ρόλο. Γιατί το θέμα είναι πότε αρχίζει. Η συνέπεια λοιπόν της αλλαγής στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα είναι μόνο για το 15, θα είναι και για το 16 και για το 17. Εξαρτάται για ποιο ταμείο. Συνεπώς αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε για το προσχέδιο προπολογισμού και παράλληλα για την αναθεώρηση του πολιτισμού δημοσιονομικού πλησίου είναι για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των πολιτικών μας κατά την συγκεκριμένη περίοδο. Πρέπει να το κάνουμε για να διευκολύνουμε τη διαδικασία. Ευχαριστούμε κύριε Ολμπρίχτ. Είναι μια κατάσταση αυτή, κάπως ιδιαίτερη γιατί όλοι θέλουμε να δώσουμε όθηση στις επενδύσεις για να έχουμε ανάπτυξη. Να λοιπόν που ένα πολιετές πλαίσιο το οποίο εγκρίθηκε στα τέλη του 2013 και ίσως αυτό να είναι το λάθος του παρελθόντος είναι ότι αργήσαμε να τον κρίνουμε. Χρειάστηκαν 18 μήνες για να καθοριστούν τα προγράμματα, οι διαδικασίες και οι κανόνες. Αυτό δείχνει την αδράνεια με την οποία λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε αυτή την αδράνεια, πρέπει κάτι να κάνουμε. Και να εκφράσουμε την επιθυμία και να πούμε ότι ό,τι δεν χρησιμοποιήθηκε το 2014 να διατεθεί το 2015 και να μετρήσει διπλά. Γιατί είναι κάπως παράδοξο να ξεκινάμε με το επενδυτικό πρόγραμμα του Juncker και οι διατάξεις που έχουμε στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να μας καθυστερούν τόσο πολύ. Τι έχετε να πείτε η Γενική Συγκήτρια, τίποτα. Ωραία. Οι τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 25 Μαρτίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών θα λάβει χώρα στις 16 Απριλίου και στην Ολομέλεια θα περάσει το θέμα στις 29 Απριλίου. Τότε θα ψηφίσουμε το διορθωτικό προπολογισμό 2 για το 2015. Έρχομαι τώρα στην κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Έχουμε την υπόθεση ΕΖΕΦ, Μωρή Ντικρό, τη Γαλλία. Ο κύριος Ντενό Όντω, η Γαλλία ζητάει να κινητοποιηθεί το Ταμείο για τι συνέπειε από την ε, παγκοσμιοποίηση. Πρόκειται για την εταιρεία Μωρή Ντικρό. Ακούστηκαν πολλά για αυτή την ε, περίπτωση. 2.395 απολύθηκαν. Και σήμερα χρειάζονται βοήθεια. Ήταν αρχικά 4.911. Η εταιρεία αυτή ήταν η δεύτερη μετά την Geodis και χρησιμοποιούσε 4.500 οχήματα κάθε μέρα. Μετά την οικονομική κρίση και την παγκόσμια κρίση, οι μεταφορές ε, αυτές μειώθηκαν κατά 13,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 21% ανάμεσα στο 2007 και το 2012 στη Γαλλία η παραγωγή στην Ευρώπη, η εξέλιξή της είχε σαν αποτέλεσμα να χειροτρέψει η κατάσταση στην Ευρώπη και να αυξηθεί και το κόστος λόγω της αύξησης τιμής ε, της βενζίνης, ε, των υλικών ε, που χρησιμοποιεί η εταιρεία κλπ. Οπότε αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση η επιχείρηση αυτή από τις 6 Νοεμβρίου και στο Μάιο του 2014 έκλεισε η επιχείρηση. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η Μωρή Global, η οποία κάλυψε κάποιες ε, περιπτώσεις, κάπου 2.500 επαναπροσέλαβε, ενώ οι υπόλοιποι έμειναν χωρίς δουλειά. 2.513 αποφάσισαν να δεχτούν την συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Η διαδικασία προχώρησε. Το γαλλικό κράτος προκατέλαβε, επειδή δεν υπήρχαν καθόλου χρήματα, το Υπουργείο Εργασίας χρηματοδότησε τη διαδικασία αυτή στην αρχή της. Καλώς. Ποιος θέλει το λόγο? Κανείς? Ευχαριστούμε κύριε Ντελανό. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 23η Μαρτίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών την 1η Απριλίου και όχι την 31η Μαρτίου, γιατί τότε έχουμε το σεμινάριό μας. Και στις 15 Απριλίου θα ψηφίσουμε στην Μίνη Ολομέλεια. Συνεχίζουμε τώρα. Και περνάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εδώ έχουμε τροποποίηση του κανονισμού. Αύξηση του ποσού της αρχής χρηματοδότησης για την απασχόληση των νέων. Είναι μια πρωτοβουλία που θα θυμόσαστε ότι άρχισε στα τέλη του 2013 και αποτέλεσε αντικείμενο διατάξεων ε, κανονισμού πολύ συγκεκριμένων γιατί η προχρηματοδότηση ήταν περιορισμένη στο 1% των προβλεπόμενων δαπανών. Συν 50% θα έλεγα, δηλαδή 1,5% συνολικά, για τις χώρες μέλη που βρίσκονται σε οικονομική αρρωγή. Η πρόταση λέει η προχρηματοδότηση αυτή να ανέβει στο 30% που είναι σημαντικό 30% υπό τον όρο ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να βάλει 50% των δαπανών μέσα στους 12 πρώτους μήνες. Αυτή είναι μια αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου οι χώρες να επιταχύνουν τη διαδικασία. Το Συμβούλιο εξάλλου είναι αυτό το οποίο εξέφρασε την επιθυμία αυτή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε έκθεση βάσει του άρθρου 53. Μου αναθέσατε και την ευθύνη να συντάξω την έκθεση αυτή. Οι παρατηρήσεις που έχω να κάνω είναι οι εξής. Προκειμένου η διάταξη αυτή να λειτουργήσει πλήρως στις ενδιαφερόμενες χώρες, είναι πολύ σημαντικό οι χώρες αυτές να προχωρήσουν στις αναγκαίες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Εξάλλου, μπορούμε να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα. Δηλαδή αν σε μια συγκεκριμένη χώρα υπάρχει ιδιαίτερη υψηλή ανεργία και τα κονδύλια αυτά οριοθετούνται γεωγραφικά, σε περιοχή που υποφέρει ιδιαίτερα από την ανεργία, 25% είναι το όριο το οποίο επιλέχθηκε. Αν λοιπόν σε αυτήν τη γεωγραφική περιοχή υπάρχει περιορισμένη απασχόληση, νέοι ναι, αυτοί θα έπρεπε να θαρρυνθούν και να μετακινηθούν σε άλλες περιφέρειες όπου οι δυνατότητες απασχόλησης είναι μεγαλύτερες. Και θέλω να υποφεληθώ από την συζήτηση αυτή για να σας πω ότι θα ήθελα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα πειραματικό δοκιμαστικό πρόγραμμα για την κατάρτιση στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει προχωρήσει πολύ με το Εράσμους για τους φοιτητές. Υπάρχουν διατάξεις από τις οποίες μπορούν να αποφεληθούν και οι μαθητευόμενοι. Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στην κινητικότητα μετακινούνται για διαμονές μερικών εβδομάδων μόνο. Οπότε θα θέλαμε να τους ενθαρρύνουμε να μετακινούνται για περισσότερο, για 6 για ένα χρόνο, σε κάποια άλλη χώρα που δεν είναι η δικιά τους. Αναφίβολα οι χώρες οι οποίες προχώρησαν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και έχουν ανταγωνιστική οικονομία είναι καλύτερα σε θέση να μειώσουν την ανεργία των νέων, ανεργία των νέων που είναι ένα σκάνδαλο. Οι χώρες λοιπόν που έχουν ε, αυτό το σύστημα της μαθητείας δίνουν ευκαιρίες στους νέους να βρουν δουλειά. Και σίγουρα σε τέτοιες χώρες μπορούν πολύ περισσότερο να βρουν δουλειά οι νέοι παρά στις άλλες χώρες. Αυτά είχα να σας πω λοιπόν, παρουσιάζοντάς σας την έκθεσή μου. Ποιος θέλει το λόγο. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη 17η Μαρτίου. Στις 24 Μαρτίου θα ψηφίσουμε. Όχι, την 1η Απριλίου θα ψηφίσουμε. Και στις 16 Απριλίου η Επιτροπή Απασχόλησης που είναι υπεύθυνη επί της ουσίας θα ψηφίσει. Η κυρία Λιάτ Νιριάιντα έχει έκθεση πρωτοβουλίας για τις ευκαιρίες ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι εδώ όμως σήμερα η συντάκτρια της γνωμοδότησης αυτής η Γκουε. Θα έχει κάποιον αντικαταστάτη. Υπάρχει κάποιος που αντικαθιστά τη συντάκτρια, την κυρία Λιάντα Νιριάντα. Πάντως ζήτησε να αρχίσει η συζήτηση ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που το επιθυμούν, α, όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. Προκειμένου όσοι θέλουν να εκφραστούν για το θέμα να μπορούν ήδη από σήμερα να το κάνουν. Θα γνωρίζετε την γνωμοδότηση αυτή, την έχετε φαντάζομαι υπόψη σας. Ποιος θέλει το λόγο λοιπόν? Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Οι τροπολογίε πρέπει να υποβληθούν το αργότερο το 19η Μαρτίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών θα λάβει χώρα την 1η Απριλίου. Α, παρακαλώ κύριε Τόρβατς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς θεωρούμε ότι ορισμένες διατυπώσεις που επιλέγει η συγγήτρια στην έκθεσή της είναι ας πούμε κάπως ασθενής. Ήρθαμε σε επαφή με το γραφείο της σήμερα για να κάνουμε κάπως πιο δεσμευτικές διατυπώσεις αυτές ή τέλος πάντων έτσι ώστε να λένε κάτι για το πρόβλημα. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Ευχαριστώ. Πρώτη Απριλίου η ψηφοφορία και η ορμένης 14 Απριλίου. Εσείς κύριε Τελανού έχετε συντάξει έκθεση για την πρόθεση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής στην Ενώση. Ήθελα να παρουσιάσω την έκθεση αυτή, κύριε Πρόεδρε, διότι είδα ποια είναι η μεγάλη σημασία των διαθετικών ταμείων στην επικράτεια της Ένωσης και θέλω να τονίσω τον ρόλο τους στην πολιτική της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. Τα ταμεία αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για την απασχόληση. Εφόσον λοιπόν, αν δεν υπήρχε μάλλον το ΦΕΝΤΕΡ και το ΕΦΕΣΥ... θα είχαμε δει σημαντικότατη μείωση των ε, ΑΕΠ και πολύ μεγαλύτερη ανεργία. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν γιατί βεβαίως πάντα υπάρχει και μια χρονική απόσταση ανάμεσα στην ανάληψη των δεσμεύσεων και στην εφαρμογή τους. Η πολιτική αυτή συνοχής συνεχίζεται σήμερα και βεβαίως αυτό είναι ικανοποιητικό. Συνεχίζεται με νέους πολιτικούς προσανατολισμούς και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη την παιδεία, την οικονομία, ε, κυρίως την εξοικονόμηση μάλλον εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακος, την ενίσχυση του ρόλου των μικρών και μεσών επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να παίξουν πραγματικά ένα ρόλο που είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη. Είναι αληθές εξάλλου ότι αυτή η νέα πολιτική συνοχής βασίζεται σε μια στρατηγική ευφυή και βιώσιμη. Και στην περιοχή της Γαλλίας από όπου έρχομαι παίζουμε το παιχνίδι αυτό διότι εξετάσαν ποιες είναι οι κατευθύνσεις, οι καλύτερες κατευθύνσεις για την περιοχή αυτή και έτσι είναι σωστό να γίνει και έφνης οι κατευθύνσεις που δίνει η συνθήκη της Ένωσης ανοίγουν προοπτικές για την μείωση των αποκλήσεων είτε κοινωνικών είτε γεωγραφικών υποστήριξη λοιπόν στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και χαιρόμεθα κιόλα που έχουμε πετύχει και την θέσπιση των περιφερειών μετάβασης που δεν έχουν φτάσει δηλαδή ακόμα σε απόλυτη ανάπτυξη αλλά αξίζει τον κόπο να ενισχυθούν και προτεραιότητα των ταμείων αυτών στη νέα πρόπτικη θα είναι να δοθεί όθηση στην ανάπτυξη στη βάση μιας ενδιαφέρουσας στρατηγικής που ζητεί να ενισχυθούν οι επενδύσεις και να συγκεντρωθεί η χρηματοδότηση σε ορισμένους τομείς προτεραιότητας όπως αυτούς που ανέφερα πριν καθώς επίσης να είναι μετρήσιμη μάλλον η επιτυχία των πολιτικών αυτών. Και ιδίως της πολιτική συνοχής, ιδίως στις πόλεις εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και σε αυτό να συνεργαστούν όλοι οι εταίροι που ενδιαφέρονται για την οικονομική, κοινωνική και ε, εδαφική ανάπτυξη και συνοχή με μεγάλο αριθμό εταίρων, με διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται. Είναι ικανοποιητική εξέλιξη αυτή και ο προϋπολογισμός μάλιστα αποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Έχω λοιπόν γνωμοδότηση η οποία βασίζεται ιδίως στην ανάγκη να φροντίσουμε ώστε το πρόγραμμα επενδύσεων που ε, προτείνει ο πρόεδρος Γιούνκερ να βασιστεί στην αρχή της προσθετικότητας, δεύτερος άξονας της εκθεσής μου είναι, όπως έχουμε πει άλλωστε εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, το θέμα που επιμένει των απλήρωτων λογαριασμών, η συνοχή και βεβαίως πρέπει να ζητήσουμε από Κομισιόν και Συμβούλιο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στον τομέα των απλήρωτων λογαριασμών και στην ανάλυση των θετικών στοιχείων της μεταρρύθμισης αρχιτεκτονικής Νομίζω πρέπει να επισημάνουμε τα νέα ε, ε, χρηματοδοτικά εργαλεία και τη στόχευση σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων, χωρίς να λησμονούμε ότι υπάρχουν εδαφικές προτεραιότητες, ε, συγγνώμη, ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν ορεινές περιοχές και ούτω καθεξής και επομένως πρέπει να δώσουμε και ένα ελάχιστο ευκαμψίας για να μπορέσουμε να μπορέσουν να αποδώσουν τα διαθωτικά ταμεία. Ε, επιμένω δε ιδίω στο ότι η ένταξη των κριτηρίων μακροοικονομικών, μακροοικονομικής αιρεσιμότητας μάλιστα, ε, είναι εντελώ απαράδεκτη. Θα πρέπει επιτέλου να μπορέσουμε να εκφράσουμε, να, να πούμε μάλλον ότι δεν πρέπει να υπάρχει μακροοικονομική αιρεσιμότητα, είναι σημαντικό και επίσης είναι σημαντικό να χωρίς να λησμονούμε τους ιδίους πόρους και τις πληρωμές. ώστε να καταλήξουμε σε υλοποίηση των ε, έργων. Ευχαριστώ πολύ για την ανάπτυξη του θέματος. Έχετε παρατηρήσει. Φερνάντης. Πολύ σύντομα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα της πολιτικής συνοχής που έχουν ήδη συζητηθεί. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατό. Πέραν αυτού, στα πλαίσια του πολιετούς ε, ε, δημοσιονομικού πλαισίου, ε, τα όσα έχουν συμφωνηθεί θα πρέπει να εφαρμοστούν και δεν πρέπει να υπάρξει καμία αμφιβολία, καμία καθυστέρηση σε σχέση με τις πληρωμές. Πέραν αυτού, ε, η πολιτική σύνοχης σε πολλά κράτη-μέλη βοηθά όχι μόνο για τις υποδομές αλλά για την ευθεία ανάπτυξη, για τις επιχειρήσεις και για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η εδαφική συνοχή προχωρά χέρι-χέρι με την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Φερνάντες, η κυρία Βάνα. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της δικής μου πολιτικής ομάδος σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη γνωμοδότηση η οποία σαφέστατα είναι θετική και αποτελεί καλή βάση για τη συζήτηση. Ιδίως συμφωνούμε με τη δήλωσή του περί της μεγάλης σημασίας της πολιτικής συνοχής, ιδίως μέσα στην κρίση, καθώς επίσης και τη σημασία των δημοσίων επενδύσεων και για την επίλυση του προβλήματος των απλήρωτων λογαριασμών και για την κριτική του βεβαίως ε, είμαστε απόλυτα σύμφωνες για την κριτική δηλαδή που κάνει στην μακροοικονομική αρεσιμότητα. Εμείς θα θέλαμε να περιλάβει και ορισμένα άλλα κέντρα βάρους που θα τα θέσουμε κι εμείς αφενός την ε, τον τονισμό της συνεργασίας και των τοπικών εταίρων και φορέων, δηλαδή της κοινωνίας των πολιτών, αυτό νομίζω ότι μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας των διαθετικών ταμείων είναι και κάτι δίτο μοναδικό. Ιδίως τώρα μάλιστα που μιλούμε για βελτίωση της εφαρμογής του σχεδίου επενδύσεων του Πρόεδρου Γιούνκερ θα πρέπει η αρχή αυτή της, ε, της συνεργασίας να έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Το ίδιο πρέπει να τονιστεί η σημασία της πράσινης οικονομίας και των πράσινων θέσεων απασχόλησης, ιδίως μέσα στην ε, πολιτική της συνοχής. Ένα σημαντικό μέρος δηλαδή των επενδύσεων αυτών θα πρέπει να κατευθυνθεί σε μέτρα πρασινίσματος της οικονομίας. Επίσης, εν ώψη των εκθέσεων του ελεγκτικού συνεδρίου, σωστό είναι να τεθεί και το θέμα της διαφάνειας, του capacity building και της λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Βρίσκω ότι αυτά τα θέματα είναι σημαντικά, θα τα περιλάβουμε σε τροπολογίες, αλλά στο σύνολο δηλώνουμε ικανοποιημένε με την πορεία της γνωμοδοτήσεως. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, λέει κύριος Ομαζή. Θα ήθελα εξ ονόματο τη πολιτική ε, μα ομάδα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ντρινανό. Είναι πολύ ε, εξαιρετική ποιότητα οι προτάσει του και θα κάνω μόνο ε, κάποιε παρατηρήσει. Στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία διαπραγματευτήκαμε όλους τους κανονισμούς σε σχέση με την πολιτική συνοχή που έχουν πλέον σταθεροποιηθεί και θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι το 2020. Εγώ μετήχα παραδείγματο χάρη στις διαπραγματεύσεις για την περιφερειακή πολιτική ε, και υπήρχαν αυστηρότατοι περιορισμοί για την μακροοικονομική ε, ρεσιμότητα. Έχουν ληφθεί πλέον οι αποφάσεις και αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι οι προοπτικές μετά το 2020. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε τώρα διότι η δεύτερη έκθεση για την συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας δείχνει ότι ειστερούμε σε σχέση με τους στόχους μας μετά την εκδήλωση της κρίσης το 2008. Και κάποιοι που επιδιώκουν με τον πολιτικό τους λόγο να αποδυναμώσουν τη μοναδική ένδειξη αλληλεγγύης, δηλαδή την πολιτική συνοχής, θα πρέπει να μας βρουν απέναντί τους όταν ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να περιοριστεί η πολιτική συνοχή σε διότι εξυπηρετείται ταυτόχρονα με την πολιτική συνοχή η αναπτυξιακή πολιτική με σημαντικότατες επενδύσεις στις ε, περιφέρειες. τίποτα δεν έχει ρυθμιστεί τελεσίδικα, ξέρουμε ότι το 2016-2017 στην ενδιάμεση αναθεώρηση ε, ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε και πάλι πρόβλημα με τις πληρωμές και στο τέλος της προγραμματικής περίοδου ενδεχομένως να μην είναι πλέον διαχειρίσιμη η κατάσταση. Εδώ θα σταματήσω εδώ διότι έχουμε ήδη ε, καθυστερήσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε νομίζω ότι όλα είναι ξεκάθαρα αυτά. Ναι, ναι, λέει ο κύριος ε, Ντενανό, αυτά περιμένα να πούνε οι συνάδελφοι και περιμένω τις ε, τροπολογίες. Ο κύριος Σαρτής συνεχίζει εκτός μικροφώνου. Εκτός μικροφώνου. Ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ. Ο Σαλ Γκέρνς, ο συνάδελφός μας, έχει καταθέσει ένα σχέδιο. Ζητά συγγνώμη διότι κολλείται και δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Ε, το σχέδιο του λοιπόν δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Ασχολείται μόνο με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ε, δεν ε, φεύγει του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Τρία είναι τα βασικότερα ζητήματα. Ζήτα στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου να λυθεί υπόψη η αύξηση των διαρθρωτικών αναγκών ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια. Θεωρώ ότι όλες οι πολιτικές ομάδες μπορούν να το δεχτούν. Επίσης, από πλευράς προϋπολογισμού και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ικανοποιητικά την αυξημένη ανάγκη για την ανθρωπιστική βοήθεια, θα πρέπει να υπερασπιστούμε την αρχή ανάμεσα, τις ισότητα ανάμεσα στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και στι πιστώσεις ε, πληρωμόνε. Συνέχεια για το αναπτυξιακό εργαλείο μας ζητά ε, να σεβαστούμε την αρχή της χρηματοδότησης του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος για την αναπτυξιακή ε, βοήθεια. Ιδού. Αυτά είναι τα τρία βασικά σημεία με τα οποία πρέπει να συμφωνήσετε ούτως ώστε να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας στον ε, κύριο Σάλ για το προσχέδιο. Ο κύριο Σαρτή, σας ευχαριστούμε που αντικαταστήσατε τον ε, κύριο Γκέρνς. Ε, το, ξέρω ότι το 0,7% είναι αμεληταίο, αλλά υπάρχουν ε, δημοσιονομικοί περιορισμοί σε επίπεδο κρατών μελών και δυσκολεύονται ακόμη και με αυτό το ποσοστό να συμμορφωθούν και μεταξύ άλλων θα μας βοηθήσει αυτό το 0,7% να αναχαιτήσουμε τα μεταναστευτικά κύματα. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στη ψηφοφορία. Για τις μεταφορές είναι ονομαστική η ψηφοφορία, σας το υπενθυμίζω. Λοιπόν, για το ε, Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, Attica Broadcasting Ελλάδα, ε, έκθεση του κύριου Κίρτσου. Είστε έτοιμοι να ψηφίσουμε στην παράγραφο 7. Μία συμβαστική α. Ποιος είναι υπέρ. Παρακαλώ, με ανάταση χειρός, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8α, τροπολογία 2. Υπέρ, εισηγητη Ποιοι είναι υπέρ? Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 8β. Τροπολογία 3. Υπέρ εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 9α. Τροπολογία 4. Υπέρ ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 9β. Τροπολογία 5. Υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 9 γάμα, τροπολογία 6 υπέρ, ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 7, παράγραφος 9. Α, καλύπτεται από τη συμβαστική α βλέπω εδώ. Παράγραφος 9, ε, τροπολογία 8 υπέρ, ο εισηγητής υπέρ. Κα, κατά αποχές 9F τροπολογία 9 υπέρ ο εισηγητής υπέρ όλοι υπέρ είστε κατά δεν υπάρχουν ούτε αποχές για το σύνολο του ε, κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται Ψήφισαν όλοι πέρας. 29 ψήφοι υπέρ, 3 κατά εγκρίνεται. Πάλι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, Άτικα, Publishing Activities. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Χριστοφόρου. Για την παράγραφο 5, η 1 υπέρ, ο εισηγητής υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7 συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 8 Παράγραφος 8α, μάλλον τροπολογία 2, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 8β, Τροπολογία 3, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν. Εγκρίνεται. Ε, 9α, τροπολογία 4, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 10α. Ε, Η 10α καλύπτεται από τη συμβαστική α 10β, η τροπολογία 6 υπέρ, ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10, ε, η τροπολογία 7 υπέρ, ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 10 δέλτα, τροπολογία 8 υπέρ, ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές δεν υπάρχουν για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε μόλις τώρα. Ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίθηκε η έκθεση με 30 ψήφους ε, υπέρ προς 3 κατά. Έκθεση για τη Lufthansa Technik. Α, ο κύριος Ντενανό, παρακαλώ. Α, να προσθέσετε την ψήφο μου γιατί δεν λειτουργούσε το μηχάνημα. Και εγώ υπέρψηφισα. Λοιπόν, Lufthansa Τεκνίκ, ο κύριος Νεγκρέσκου είναι ο εισηγητής, παράγραφος 1, τροπολογία 2, υπέρ εισηγητής υπέρ. Κατά. Ε, δεν είμαι σίγουρος, ονομαστική ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. Ναι, εγκρίθηκε 17 προς 16. Όντως, δεν ήταν ε, σίγουρο. Ε, τροπολογία είναι υπέρ, υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αποχές τις ξέχασα. Εγκρίνεται. Ε, παράγραφος τροπολογία 4, υπέρ, ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Έλεγχο ζητάτε εξακρίβωση. Τροπολογία 3, με, με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίσαμε την 1, την, 3 με ανάταση χειρός και μου φάνηκε ότι υπήρχε πλειοψηφία για να εγκριθεί. Η τροπολογία 1 είναι στο τέλος. Το 1 είναι στην αρχή. Ε, ε, το ένα είναι στο τέλος. Συγγνώμη, αλλά ο κατάλογος ψηφοφορίας των σοσιαλιστών άρχιζε από την τροπολογία 1 και ακολουθήσαμε τον κατάλογο, δεν σας ακούσαμε όταν εκφωνούσατε την, τον αριθμό της τροπολογίας και ψηφίσαμε βάσει της δικής μας λίστας. Ε, εξού και το πρόβλημα για την τροπολογία 2 είναι υπέρ φυσικά γιατί είναι του εισηγητή μας, καταλαβαίνετε. Τέλος κατά τύχη ψηφίσατε σωστά. Εν Τροπολογία 3 και εσείς νομίζατε είναι η 2 ή 3. Αυτό έγινε. Τώρα το ψηφίσαμε όμως. Ε, τροπολογία 4 την ψηφίσαμε. Τροπολογία 5 παραγράφος 6-1 υπέρ ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 6-1 ε, τροπολογία 6 υπέρ ο εισηγητής υπέρ. τροπολογια 6 υπερ ο Αποχές Εγκρίθηκε. 7. Η τροπολογία 7 υπέρ, ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν. Εγκρίνεται 7. Β. Τα τροπολογία 8 υπέρ, ο υπερ υπέρ. Κατά. Όχι, αποχές ούτε. Εγκρίνεται. 8-1 τροπολογία 9 υπέρ, ο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 8β, τροπολογία 10, υπέρ, ο εισηγητής υπέρ. Κατά, αποχές, κανείς. Ε, εγκρίθηκε Σ. τροπολογία 11, υπέρ, ο εισηγητής υπέρ. Κατά, όχι, ούτε αποχές, εγκρίνεται. Ε, η 9-1, τροπολογία 2, υπέρ, ο εισηγητής υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10, η τροπολογία 13, ε, ε, υπέρ, της υπέρ. Κατά. Ε, έλεγχος. Ηλεκτρονικός. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 10α, ε, τροπολογία 14. Είναι υπέρ ο εισηγητής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Εκτιμώντας D, τροπολογία 1. Κατά ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. περίφθει 15 προς 17. Και για το σύνολο του σχεδίου... Ε, ζητώ συγγνώμη, λέει η κυρία Γκαρδιά Σαβάλα. Ε, δεδομένου ότι κάναμε αυτό το λάθος θα σας ζητήσω από σας Πρόεδρε και τους συναδέλφους να, ξαναψηφίσουμε την τροπολογία 3. Χωσή Μανουέλ, τι κάναμε λάθος. Νομίζαμε ότι ψηφίζαμε άλλη τροπολογία. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τροπολογία 3. Εγκρίθηκε. Ε, από ό,τι θυμάμαι. Εγκρίθηκε έτσι δεν είναι. Για το σύνολο το κειμένου όπως τροποποιήθηκε ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Πέρας. Εγκρίθηκε. 28 ψήφοι προς 5. Κυρία Γκόρδια Ζαμπάλ, για τον προπολογισμό 2015 έχουμε τρεις εκθέσεις για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, ε, ψηφοφορία για τη μεταφορά, με νομαστική ψηφοφορία. Αν επιτρέπετε να ψηφίσουμε ομού για τις τρεις μεταφορές. Ωραία. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Όχι. Ναι. Πέρας τώρα. Υπερψηφίστηκαν 30 ψήφοι προς 3. Για τα υπόλοιπα τμήματα δεν υπάρχει κανένα αίτημα ούτε για την κτηριακή πολιτική. Ολοκληρώνουμε την ημερήσια διάταξη. Υπό τα διάφορα υπάρχει κάτι. Όχι. Λήξη. Παρακαλούνται οι συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα. Διότι θα συνεδριάσουμε.